Συνάδελφοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Ας συνεχίσουμε. Έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα όλη μέρα, έχουμε και συντονιστές το μεσημέρι. Όμως, έχουμε να εξετάσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ακούσουμε δηλαδή τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Γνωρίζουμε πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτή τη Επιτροπή, ιδιαίτερα θέματα ασύλου και μετανάστευση ε, που σχετίζονται με την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Μια κατάσταση που είναι δυσβάσταχτη, όπω γνωρίζουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε την ε, τις εξελίξεις για τους ε, φακέλους που αφορούν το Δουβλίνο και τη σχέση που υπάρχει με την Ελλάδα και το μπλοκάρισμα του κανονισμού του Δουβλίνου στο Συμβούλιο. Καθώς και το πώς όλο αυτό επηρεάζει το σύστημα ασύλου. Όπως θα γνωρίζετε, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Η στήριξη που λαμβάνει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορώ ε, απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Έχουν συζητηθεί οι συνθήκες υποδοχής, τα κονδύλια, οι βιώσιμες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του ασύλου και της μετανάστευσης και οι σχέσεις ε, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν την ε, ώρα που έρχεται για όλα αυτά και για ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Υπουργό, κύριο Χρυσοχοίδη. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραβρεθώ σήμερα στην συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Το θεωρώ εξαιρετική τιμή και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για έναν ειλικρινή, ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα χωρίς εισαγωγή. Η χώρα μου, η Ελλάδα, η οποία αποτελεί το ανατολικό μεσογειακό σύνορο της Ευρώπης, αποτελεί σήμερα το σημείο εισόδου χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων που προέρχονται από την Ασία αναζητώντας μια καινούργια ζωή στην Ευρώπη. Η είσοδος γίνεται από τη θάλασσα και η εκκίνησή τους γίνεται από τη γειτονική χώρα την Τουρκία και εδώ χρειάζεται να διευκρινίσω ότι η απόσταση μεταξύ της τουρκικής, των τουρκικών ακτών και των ελληνικών νησιών, συγκεκριμένα της Λέσβου, της Άμμου, της Κό και άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα σε 13 περίπου λεπτά με, μια, με ένα ταχύπλο φουσκωτό, μια ταχύπλο βάρκα να καταφθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα στις ακτές των ελληνικών νησιών. Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εντάσσεται στην κοινή δήλωση των δύο μερών εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου από τον Μάρτιο του 2016 η Τουρκία εισπράττει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια για την διαχείριση των τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενεί στο έδαφος της από τη Συρία με ταυτόχρονη υποχρέωσή της να ελέγχει τα σύνορα προς την Ευρώπη και να δέχεται επιστροφές από τα ελληνικά νησιά όσων δεν υπάγονται σε διεθνή προστασία πάντα σύμφωνα με το γράμμα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή είναι με δύο λόγια η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το Μάρτιο του 19, του 16 με συγχωρείτε, η οποία είναι σε ισχύ σήμερα. Οι ροές μέχρι τον Ιούλιο του 2019, εδώ και λίγους μήνες δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν διαχειρίσιμες. Από τον Αύγουστο οι ροές αυξήθηκαν περίπου 120%. Με αποτέλεσμα να φτάνουν κάθε μέρα με βάρκες οι άνθρωποι μέχρι τον αριθμό και χίλια άτομα κάθε μέρα στα νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου. Και πρωτίστως θα έλεγα στη Λέσβο. Το πρόβλημα στα νησιά είναι εκρηκτικό. Έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα διαχείρισης, ακόμα μπορώ να σας πω ότι ακόμα κι αν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της logistics ε, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Γιατί σκεφτείτε, αναλογιστείτε πόσους ανθρώπους μπορεί να εξετάσει ένας γιατρός τη μέρα. Πόσους μπορεί να καταγράψει ένας υπάλληλος τη μέρα πόσους μπορεί να δακτυλοσκοπήσει κανείς σε μια μέρα όταν την επόμενη μέρα έρχονται άλλοι 500. Μόνο στο ένα νησί. Είναι αδύνατον να υπάρξει συνθήκη φιλοξενίας σε ανθρώπινο επίπεδο με αυτούς τους ρυθμούς και αυτούς τους πληθυσμούς που καταφθάνουν κάθε μέρα στα ελληνικά νησιά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή ένας όλεθρος ένας κοινωνικός όλεθρος. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα με αξιοπρέπεια μόνη της χωρίς καμιά συνδρομή προσπαθεί να διαχειριστεί αυτήν την ανθρώπινη πλημμύρα. Γίνεται λόγος πολλές φορές για ένα καράβι που μεταφέρει 100-200 ανθρώπους από τη Λιβύη προς την κεντρική, στην κεντρική Μεσόγειο και γίνεται συζήτηση για να υπάρξει μια κατανομή αυτών των ατόμων. Εδώ σας ε, αναφέρω νούμερα, μεγέθη, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με κανένα σημείο της ε, Μεσογείου. Να σας δώσω επίσης ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μεταφέρθηκαν από τα νησιά, κυρίως από τη Σάμο, περίπου 4.000 άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας για να αποσυμφορήσουμε τα νησιά γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας. Η αποσυμφόρηση των νησιών, η μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλή σημεία στην υπηρετική Ελλάδα και έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες καταγραφής τους και οι διαδικασίες για τους ετούντες άσυλο. Έφυγαν λοιπόν από τη Σάμο περίπου 4.000 άνθρωποι και ταυτόχρονα σε δύο εβδομάδες κατέφθασαν 3.000 εν τω μεταξύ. Η νέα ελληνική κυβέρνηση ψήφισε πριν από λίγες μέρες το νέο νόμο για την παροχή διεθνούς προστασίας και δρομολογεί δράσεις για την εφαρμογή αυτού του, του νόμου με στόχο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ασύλου να μη στηβάζονται οι άνθρωποι στα νησιά σε συνθήκες άθλιες και απάνθρωπες να εγγυηθεί τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και να επιστρέψει πίσω στην Τουρκία με βάση τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όσοι με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κριτήρια του νόμου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τη διεθνή προστασία. Ο νόμος αποτελεί πιστή μεταφορά της οδηγίας και των κανονισμών που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόλυτο σεβασμό στο αξιακό πλαίσιο της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Γενέβης και το ενωσιακό δίκαιο. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μία σε δύο ζητήματα. Το ζήτημα της μετανάστευσης δεν αποτελεί πρόβλημα ή πολιτικό ζήτημα ή διακύβευμα αυτών που βρίσκονται μόνο στο front line της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα το οποίο τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Και είναι ένα κεντρικό πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Και κατά ανάγκη θα αποτελεί ένα ζήτημα πολιτικής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης σε καθημερινή βάση. Και κατά ανάγκη θα υπάρξουν και συγκλήσεις και αποκλήσεις και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις προσεγγίσεις του, καθενούς ωστόσο το φαινόμενο που παρατηρείται ορισμένοι να θεωρούν εννοώ από εμά από τα μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης να θεωρούν ότι κλείνοντας τα σύνορά τους είναι ασφαλείς και ότι δεν θα επιτρέψουν αυτές τις ροές των ανθρώπων να εισέρχονται στην επικράτειά τους αυτό είναι τοπικό. Είναι υψίστη ουτοπία και ψευδέστηση. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Δεν θα επικαλεστώ την αλληλεγγύη ως έννοια που πρέπει να διακρίνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επικαλούμε τους κανόνες, το δίκαιο. Ότι όλη αυτή η Ένωση, όλος αυτός ο οργανισμός είναι κάτω από ορισμένους κανόνες, έχει χτιστεί. Οι οποίοι υποθέτω ότι πρέπει να εφαρμόζονται. Εδώ λοιπόν έχει ανατεθεί στον εθελοντισμό η εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό νομίζω δεν προάγει την Ένωση συνολικά. Είναι τοπικό επαναλαμβάνω, να πιστεύουν ορισμένοι ότι κλείνοντας τα σύνορά τους, γυρνώντας ουσιαστικά την πλάτη στο πρόβλημα ή λαϊκίζοντας, θα επιχειρήσουν να ξεφύγουν από αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο, για να τελειώσω ζήτημα, έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά ως υπουργό, παίρνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίε και θέλω να σας τις ανακοινώσω, να σας κάνω γνωστές γιατί θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πρόκειται για το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι σε δομές οι οποίες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι στην Ευρώπη. δεν είναι δομές οι οποίες τιμούν την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν με επιστολή μου στους ε, ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπόλοιπους 27 εννοώ, να πάρει κάθε χώρα εθελοντικά ένα αριθμό παιδιών. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά ανταπόκριση πλην ελαχίστων, σχεδόν ενός. Και δεν είναι ζήτημα πια ούτε αλληλεγγύης πια αυτό ούτε κανόνων. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Είναι ζήτημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού πώς αντιλαμβάνεται την περίθαλψη, την προστατευτική φύλαξη και το μέλλον αυτού του αριθμού των παιδιών. Επικαλούμε λοιπόν την ευαισθησία σας, επικαλούμε την ε, δυνατότητά σας να κινητοποιήσουμε όλες τις κυβερνήσεις, να κινητοποιήσουμε όλη την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε ένας μικρός αριθμός σε κάθε χώρα να φιλοξενηθεί και να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τα ανήλικα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Now, the usual round... Σας ευχαριστούμε. Thank you. Thank you for your testimony. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μαρτυρία. Ήταν καθηλωτική πραγματικά. Ακούσαμε λοιπόν από τον Έλληνα Υπουργό για αυτό το θέμα, τα προβλήματα στην μετανάστευση και στο άσυλο ήταν μια πραγματικά καθηλωτική μαρτυρία, έγινε έκκληση για αλληλεγγύη. Εδώ και 10 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 80, οφείλουμε να αναλάβουμε δράση. Η νομοθεσία είναι δεσμευτική για όλους για τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Θα περάσουμε στον γύρο των ερωτήσεων. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές για δύο λεπτά και έπειτα θα έχουμε λίγο χρόνο, ένα λεπτό καθένας για τα μέλη της Επιτροπής. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε φορτωμένη μέρη σε διάταξη και δεν πρέπει να καθυστερούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον συντονιστή του ΕΛΚ, ο κύριος Λένερς. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, ειλικρινή αξιολόγηση της ε, κατάστασης στην Ελλάδα. Εκπροσωπείτε την ε, νέα κυβέρνηση της Ελλάδας, γι' αυτό θα ήταν άδικο να περιμένουμε θαύματα, αλλά αυτό συμβαίνει τελευταία. Θαύματα περιμένουμε. Οι τελευταίοι μήνε ε, της κυβέρνηση έχουν δείξει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, στρατηγική, εθνική για την ε, υποδοχή των ε, μεταναστών με βάση το νομικό πλαίσιο για την πιο αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων και των επιστροφών. Το επόμενο έτος αναμένεται να μεταφερθούν 20.000 ε, πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα. Έχουμε παρατηρήσει αύξηση των ε, εισόδων ε, ανθρώπων οι οποίοι πολλές φορές δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου από την ε, στιγμή της θέσης ισχύ της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες, υπάρχουν και δυσκολίες για τα ελληνικά νησιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ακούμε αρκετές κριτικές και ζητούνται βιώσιμες λύσεις. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν κατευχήν, γι' αυτό λοιπόν εσείς γιατί θεωρείτε πως ε, υπάρχουν προβλήματα και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Έπειτα, αυτές οι 20.000 ανθρώπων που θα μεταφερθούν από τα νησιά ε, είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται χειμώνα. Σε ποια βήματα γίνονται από την ελληνική πλευρά για να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής στα νησιά και τον χειμώνα. Τέλος, αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη Είπατε σαφέστατα ότι η μετανάστευση αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η αλληλεγγύη είναι αρχή που πρέπει να ακολουθείτε και ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φαίνεται πως η έννοια της αλληλεγγύης έχει εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή από το προσκήνιο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη, να αναλυφθούν ευθύνε από όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μωράης έχει το λόγο εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η κυρία Ζήπελ λείπει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ειλικρινή εκτίμηση της ε, κατάστασης. Όλοι οι υπουργοί που έχουν έρθει από την ελληνική κυβέρνηση και εσείς και οι προκατοχοί σας είχαν έναν ανοιχτό διάλογο με την Επιτροπή αυτή και εκτιμούμε απόλυτα αυτό που κάνετε. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και είμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση όταν κάνουμε ερωτήσεις, όταν κάνουμε ερωτήσεις σε υπουργούς για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση στη Μόρια, για το τι γίνεται με τις μεταφορές. Η ερώτησή μου θα είναι παρόμοια με εκείνη του συναδέλφου από το ΕΛΚ. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στο τι πρόκειται να γίνει. Αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη, όμως αυτό είναι ένα θέμα που παραμένει, επιμένει, υπάρχουν προβλήματα. Έχουν ζητηθεί από άλλες χώρες να υποδεχτούν ασυνόδευτους ανήλικους. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ορισμένοι από εμά που έχουν επισκεφτεί τη Μόρια ξέρουν πώς είναι η κατάσταση εκεί και βλέπουμε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μόρια είναι το μέρος που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση προσφύγων. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα άσχημα, ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια αυτή τη στιγμή είναι τόσο άσχημες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ακραίες. στο Συμβούλιο όταν γίνονται συζητήσεις για το πώ θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι άνευ προηγουμένου, είναι ανήκουστο το πρόβλημα, υπάρχουν ιατρικά, ε, ιατρική ανάγκη, ιατρικά προβλήματα, υπάρχουν παιδιά που δεν ε, έχουν εκπαίδευση. Είναι λοιπόν άνευ προηγουμένου η κατάσταση στη Μόρια και όσοι από εμά την ε, παρακολουθούμε ανησυχούμε πάρα πολύ. Ε, ανησυχούμε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το γεγονός ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Εσείς τι μας συστήνετε, πώς εμείς πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο για να τους ζητήσουμε να ασχοληθούν με αυτό το πρόβλημα. Και ε, τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την ελληνική νομοθεσία, δεν θέλω να ασκήσω κριτική, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς η νέα νομοθεσία για το άσυλο θα βοηθήσει την κατάσταση. Ε, μετά από τα όσα είδα βλέπω ότι θα δυσχεράνει λίγο την ε, κατάσταση. Τι, πώς νομίζετε λοιπόν εσείς ότι ε, θα βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιντφέλντ. Για το Ρινιού. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει αφαιθεί ουσιαστικά μόνη της τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει τις εισρωές μεταναστών και όλοι ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα η Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άχθος για τους ε, ντόπιου πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν έχουν παραπονεθεί σε αντίθεση με πληθυσμού σε άλλε χώρε ε, που έχουν παραπονεθεί για καταστάσει πολύ λιγότερο δραματικέ. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό που κάνετε έκκληση σε άλλα κράτη-μέλη για βοήθεια και τελικά μόνο ένα σα απάντησε πέρα από τις πολιτικές οικογένειες τι οποίες ανήκουν οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ντρέπονται βαθιά για τον, εαυτό, για τους και λυπάμαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση τόσα χρόνια τώρα είναι πραγματικά ντροπιαστικό Βέβαια σας υποστηρίζουμε και σας και τον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό δεν ε, απαλά στην Ελλάδα από τις ε, ηθικές και άλλες υποχρεώσεις της. Δεν έχω εξετάσει ακόμη λεπτομερό την νομοθεσία, αλλά δεν είναι σαφέ σε μένα πώ ακριβώ η νομοθεσία θα βελτιώσει την κατάσταση. Γιατί ουσιαστικά οι εφέσει θα γίνουν πολύ πιο δύσκολε. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν θα υπάρχει πλέον παρουσία στο πάνελ ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Πώς αυτό λοιπόν θα βελτιώσει τη διαδικασία. Και ανησυχώ που ακούω ότι υπό την νέα νομοθεσία θα έχουμε προσωπικό της αστυνομίας και του στρατού που θα επεξεργάζονται τις αιτήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ή αν θεωρείτε ότι είναι ορθό, θα ήθελα να κατανοήσω πώς θα διασφαλίσετε ότι θα έχουν την κατάλληλη κατάρταση και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν είναι αρμόδιοι υπάλληλοι μετανάστευσης, έχουν ένα διαφορετικό ρόλο και έχουν και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να με ενημερώσετε λίγο για αυτή την νομοθεσία. Και επίσης θέλω να απαντήσω στο σχόλιο του συναδέλφου από το ΕΛΚ που είπε ότι δεν ε, υπάρχουν ε, ρεαλιστικές ε, εναλλακτικέ λύσεις στη δήλωση Τουρκίας. Ναι, υπάρχει, όπως προβλέπετε από τη συνθήκη τα τελευταία 20 χρόνια, είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή ρεαλιστική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου για τους Πλασίνους, συνάδελφος ε, κυρία Στρίκ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό ε, μας παρουσίασε τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και υποστηρίζουμε πλέον την έκκλησή του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν ελεγγύη και να αναλάβουν μέρος της ευθύνης, γιατί πιστεύουμε ότι είναι εντελώς άδικο η Ελλάδα να αφήνεται μόνη της. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Εμεί θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια που μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επιμερισμό τη ευθύνη και δεν θα την αναλαμβάνει μόνο η Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμω, αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση στο να περιορίζεται τα δικαιώματα των ετούντων ασύλου. Επό την έννοια αυτή, ανησυχούμε πάρα πολύ για την νομοθεσία που υφητήθηκε και αναφερθήκατε κι εσείς. Θα αναφέρω κάποιους περιορισμούς ε, μόνο που μας ανησυχούν ιδιαίτερα, ότι περιορίζεται ο χρόνος για την κατάθεση της αίτησης, αυξάνεται η χρήση τη διαδικασία παραδεκτότητα ε, και ότι ο στρατό και η αστυνομία θα υλοποιούν τι συνεντεύξει, περιορισμοί στην πρόσβαση, αγορά εργασία, ε, στην υγεία και αυτόματα θα άρεται η προσφυγή αν ε, υπάρχει κράτηση και επίσης ε, ότι δεν ε, θα υπάρχει αναγνώριση της ευαλωτότητας για κάποιους ανθρώπους και επίσης τα θύματα που έχουν υποστεί βασανιστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό για να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, ενώ τώρα απαιτείται να ε, εξεταστούν από δημόσια νοσοκομεία και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορείτε λοιπόν να μας ε, αποξαφινίσετε λίγο την κατάσταση αυτή και πώς όλες αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με την οδηγία ε, συνδικών υποδοχής και με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Μία άλλη ερώτηση είναι ο κατάλογο για τι ασφαλεί τρίτε χώρε. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι στον κατάλογο. Υπάρχουν και άλλε χώρε στον κατάλογο. Και μπορεί ο Υπουργό να μας διαβεβαιώσει ότι θα εξακολουθούμε να έχουμε μεμονωμένη αξιολόγηση ε, των ισχυρισμών τους. Μια άλλη ερώτηση αφορά τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι η Frontex δεν έχει πρόσβαση εκεί, ότι δεν ε, επιχειρεί εκεί. Και η ερώτησή μου ε, οφείλεται το ότι υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί για αποθήσεις από την Ελλάδα στην Τουρκία. Δεν βλέπω τον κύριο Τερντίνο. Κύριο Κόφα, παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αφού άκουσα τις ερωτήσεις ε, και τα σχόλια στη συζήτηση, μπορώ να πω ότι η μόνη ρεαλιστική και ανθρώπινη λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να εισάγουμε το μοντέλο της Αυστραλίας. Δηλαδή να έχουμε εντελώ ασφαλή σύνορα και τα εξωτερικά μας σύνορα είναι τόσο ασφαλή έτσι ώστε να μην μπορούν να τα περάσουν. Δεν θα πρέπει απλώς να προβαίνουμε σε ένα διανομή, δεν θα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορούν να περάσουν τα σύνορα οι άνθρωποι με την ελπίδα ότι θα μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη για πάντα. Δεν λειτουργεί αυτό, δεν θα λειτουργήσει. Το πιο ανθρώπινο μοντέλο που θα σταματήσει τις δηλεύσεις στη Μεσόγειο και θα διασφαλίσει ότι δεν θα έχουν κέρδη διακινητές είναι απλώς να κλείσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τους ανθρώπους στις γειτονικές περιοχές έτσι ώστε να ζουν εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη στις χώρες τους. Νομίζω ότι ε, είχε δίκιο ε, ο Πρωθυπουργό ο κ. Σελβίνη. Ο ο κ. Σελβίνη όταν έκλεισε τα λιμάνια στην Ιταλία. Το συμπέρασμά μου είναι ότι αμφιβάλλω αν αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λύσει ποτέ τα πραγματικά προβλήματα αντιθέτως έχουν ε, πληρώσει αυτόν τον απαταιώνα τον Ερντογάν ε, και έχουν ξοδέψει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, και αυτός απειλεί να στείλει εκατομμύρια μετανάστες στην πυρό μα. Αυτό δεν είναι καλό και θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Επόμενο μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Προκατσίνη. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την ελληνική κυβέρνηση. Είμαι Ιταλός και η Ιταλία όπως και η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει αφαιρεθεί μόνη της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση. Σημερίζομαι την επιλογή να εγκριθεί ένας νόμος που επιταχύνει τις διαδικασίες. Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει με τη διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Περιμένετε ένα λεπτάκι να φτιάξουμε το σύστημα. Εντάξει. Ρυθμίστηκαν όλα, όχι. δοκιμάσω. Μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, λοιπόν να σταματήσει κάπως η χρονομέτρηση λόγω της καθυστέρησης. Δεν συμφωνώ όμως όταν θεωρείται ε, ουτοπιστικό το κλείσιμο των συνόρων. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση η διακυβέρνηση μετανάστασης μέσω αυστηρών, αυστηρού ελέγχου των συνόρων είναι η μόνη ρεαλιστική λύση ε, ακόμα και για μεσύντομη περίοδο αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική όμως η ανακατανομή των μεταναστών στην Ευρώπη που κανένας δεν θέλει. Το αστέκι της συμφωνίας της Μάλτας μας το δείχνει αυτό, που έγινε εδώ και κάποιες μέρες. Πολύ συχνά καταλήγει στο να καταστρέφει τη ζωή των μεταναστών αυτή η λύση, πέρα από την αποσταθεροποίηση της τάξης και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών εθνών. Αυτό που με δυσαρεστεί εμένα και το επαναλαμβάνω κάθε φορά που μπορώ, είναι ότι ποτέ δεν μιλάμε για τα αίτια της μετανάστευσης. Υπάρχει τέλεια διαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των αιτίων της μετανάστευσης. Και αυτό είναι απάνθρωπο διοντολογικά και μειοπικό σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, ο κ. Σαρβανίτης, για την ΚΟΕ, είχε το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ και ενημερώνετε το σώμα σε μια επιτροπή που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Το μικρόφωνο σας. Παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Μόνο το σεβασμό θα ήθελα να σας πω ότι οι άνθρωποι δεν είναι τσουνάμι όπως αναφέρατε στην ε, εισήγησή σας. Οι άνθρωποι είναι, έχουν όνομα, έχουν επώνυμο, έχουν και δικαιώματα φαντάζομαι ότι είναι λάθος, εκ παραδρομή. Το σημειώνω. Όμω κύριε Υπουργέ, βρίσκεται ήδη σε ισχύ ο νέο νόμο τη κυβέρνησή σα. Και συμφωνώ απολύτω με τι ερωτήσει που έκαναν οι συνάδελφοι από του σοσιαλιστέ, από το Ρινιού και από του Πρασίνου, Είμαι ακριβώ στην ίδια λογική. Γι' αυτό λοιπόν το μαζεύω. Διεθνεί οργανισμοί κύρου κατέγγυλαν πριν λίγε ημέρε στην Αθήνα τη φιλοσοφία του νέου νόμου. Μιλώ για τη Διεθνή Αμνηστία του γιατρού χωρί σύνορα, την Human Rights 360, ότι συγκρούεται δηλαδή με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να ρωτήσω για αυτό το νόμο που καταθέσατε, κύριε Χρυσοχοίδη, με ποιου ακριβώ διαβουλευτήκατε. Με την Κομισιόν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι διεθνείς οργανώσει. γιατί στην Ελλάδα δεν έγινε διαβούλευση. Σε πέντε μέρε περάσατε το νομοσχέδιο. Δεύτερο. Η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική και η υποβάθμιση του ή μάλλον η υπαγωγή του σε Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο της Αστυνομίας καθιστά το θέμα για σας από ό,τι φαίνεται θέμα βασικά ασφάλειας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά το πρόβλημα για την κυβέρνησή σας προέσχεστε και από τους σοσιαλιστές και έχει ενδιαφέρον για μένα η απάντησή σας. Είναι μεταναστευτικό ή προσφυγικό. Τι ακριβώς είναι. Και κλείνω διότι χθε ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι θα επιστραφούν μέχρι το τέλος του 2020 περίπου 10.000 άνθρωποι. Πού, κύριε Υπουργέ, σε ποιες χώρες έχετε κάνει διμερεί συμφωνίες με κάποιους που θα ήταν καλό το σώμα να γνωρίζει. Κύριε Υπουργέ, στα δέκα δεύτερα που έχω. Ακούω στελέχη σας να λένε ότι το δόγμα σας είναι να κάνουμε στους πρόσφυγες τη ζωή τους πιο δύσκολη. Αποδεικνύεται πάντως προς το παρόν ότι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. 5.000 άνθρωποι ήταν σε απαράδεκτη για μας κατάσταση στη Μόρια, επί ΣΥΡΙΖΑ, και προχθές που πήγαμε με συνάδελφό μου από την ΚΟΕ ήταν ήδη 14.000 και σήμερα μπορεί να είναι 17.000. Δεν είχατε σχέδιο κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς. Thank you. Ευχαριστώ. Ο Υπουργό έχει ένα δεκάλεπτο να απαντήσει. Προτείνω πρώτα να τελειώσει ο γύρο των ερωτήσεων, των ομιλητών που ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό το πολύ ο καθένας. Διότι ε, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, πολύ έντονο. Τέσσερους φιλοξενούμενους ομιλητές έχουμε. Έχουμε το Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον κύριο Φλάχερτη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ένα λεπτό αν έχετε ο καθένας, μετά θα έχει δέκα λεπτά ο Υπουργός και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με κάποια καθυστέρηση, αλλά όχι μεγάλη. Η κυρία Ματσόλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε εδώ σήμερα. Προσβλέπουμε σε συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί σας, όπως είχαμε ειλικρινά συνεργασία και με προκατόχους σας άλλων πολιτικών ομάδων, διότι η ομάδα μου εδώ ε, δείχνει μεγάλη κατανόηση όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η ερώτησή μου εστιάζεται περισσότερο στην επιτόπια κατάσταση στα νησιά. Οι αριθμοί που μαθαίνουμε είναι άκρο ανησυχητικοί. Περίπου 31.000 ανθρώπους στα hot spots και τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής έχουν σχεδιαστεί για το πολύ 8.000 ανθρώπους. Αν αυτό το συγκρίνεται με την κατάσταση που επικρατεί στον τη συμφωνία με την Τουρκία και τις επιστροφές, πώς σχεδιάζεται να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας στους υπουργούς στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εκπροσωπείτε μία χώρα όπου υποφέρει σαφώς δυσανάλογο βάρος αφήξεων και έχει μείνει μόνη της η χώρα σας για να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πώς θα παρουσιάσετε την κατάσταση στους συναδέλφους σας. Ένα λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Οι ειδήσει που παίρνουμε από την Ελλάδα είναι πάντα πιο ανησυχητικέ λόγω τη επιτυχημένη με συμφωνίες που έχουμε με την Τουρκία παραμένουμε παγιδευμένοι στα νησιά σε, υπερπληθυ... σε κατάσταση υπερπληθυσμού και σε απέσιες συνθήκε. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί ακόμα όσον αφορά την νομοθεσία για τη εθνή προστασία που εγκρίθηκε τι 31 Οκτωβρίου, που αποδυναμώνει το σύστημα τη αναγνώριση και προστασία των ευάλωτων στοιχείων και καθιστά πιο δύσκολη την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, αφήνοντα μεγάλο διοικητικό άχθος στον ετούντα άσυλο. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει αυτό το νόμο τόσο ώστε να μην αποδυναμώνει το σύστημα προστασίας και υποδοχής. Τι προτίθεστε να κάνετε για να εγγυηθείτε συνθήκες αξιοπρεπής ζωής στα στατόπεδα εν ώψη και του χειμώνα. Μπορείτε να εγγυηθείτε την πρόσβαση στη θεραπεία, στην παιδεία, στους ετούντες άσυλο. Και στο τέλος σας ρωτώ, πώς επιλέξατε το Υπουργείο της Μετανάστευσης να το εντάξετε στο Υπουργείο σας της Προστασίας των Πολιτών. Αυτό δημιουργεί κάποια σύγχυση, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Σασμάνη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Ε, τέσσερα χρόνια τώρα, τέσσερα χρόνια συζητάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στα εθνικά μας κοινοβούλια κουβεντιάζουμε την καπέσια κατάσταση, την πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά, στα κέντρα υποδοχής και τον αργό ρυθμό των διοικητικών διαδικασιών. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά, δεν καταλαβαίνω που το συζητάμε αυτό όταν έρχεται ο χειμώνα. Τυπικά αυτό γίνεται. Κάθε φορά που έρχεται ο χειμώνα, πιάνουμε αυτή την κουβέντα. Και τι θα κάνουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, έχετε και αιτήματα που απευθύνεται στα άλλα κράτη-μέλη και το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Όταν δούμε τι έγινε στο παρελθόν, είσαστε νέο εκπρόσωπο τη νέα κυβέρνηση βέβαια, όταν βλέπουμε τι έγινε στο παρελθόν οικονομική βοήθεια, επιχειρησιακή ε, βοήθεια δεν αμφισβητήθηκε. Λοιπόν, γιατί, για, γιατί δεν βελτιώθηκαν, η, βελτιώθηκε η κατάσταση για την επεξεργασία των ετοιμάτων. Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε, τι δράση θα αναλάβετε για να βελτιώσετε την κατάσταση ελληνικά ε, νησιά. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάρκχαρτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στη Λέσβο την περασμένη εβδομάδα, είδα τη Μόρια και από το 2015 υπάρχει χορτικότητα περίπου 3.000 ατόμων. Τώρα έχουμε πάνω από 15.000 εκεί. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι χρειάζεστε στήριξη και την έχετε ζητήσει, όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι από το 2015 δεν έχει σημειωθεί αύξηση χορτικότητα στη Μόρια. Υπάρχουν άτομα που, χιλιάδες άτομα που μένουν σε σκηνές χωρίς θέρμανση και πρέπει να περάσουν το χειμώνα σε άθλιες συνθήκες και πάλι θα έχουμε θανάτους το χειμώνα, πάλι θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό θέλω να ρωτήσω και να πω επίσης ε, ότι δεν ξέρω αν ε, πρέπει να μιλάμε για τσουνάμι και για φυσικές καταστροφές όταν πρόκειται για ανθρώπους. Ε, θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να μιλάμε για ανθρώπους και όχι για φυσικές καταστροφές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναγνωρίσω καταρχάς το έργο της ΥΠΑ ε, της ε, Αρμοστίας. Στην πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα η κατάσταση περιγράφηκε ως εκρηκτική. Αναφέρθηκε η έλλειψη ιατρικής φροντίδας, αναφέρθηκαν τεράστιες ουρές που σχηματίζουν οι άνθρωποι για νερό, για φαγητό, για να πάνε στην τουαλέτα. Υπάρχουν προβλήματα που χρήζουν άμεση ανταπόκριση και αφορούν όλους μας. Και φυσικά η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι στη ρίζα αυτού του προβλήματος. Θα ήθελα λοιπόν, μια που είστε εδώ, να σας ε, ρωτήσω ορισμένα πράγματα για τη νέα νομοθεσία για το άσυλο. Η Κομισιόν είπε ότι η νομοθεσία αυτή ε, γύρει ε, διάφορα ερωτήματα από την σκοπιά των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου. Λέτε όμως με τη νέα νομοθεσία έχουν αλλάξει τα κριτήρια αυτά. Τι έχετε λοιπόν να πείτε γι' αυτό, για, την, για τους αυστηρότερους ελέγχους και σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους Ανήλικου. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια ήταν η χώρα αυτή που σα απάντησε θετικά και ε, σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και τις μετακινήσεις στην ενδοχώρα. Από ό,τι ακούω η κατάσταση έχει επιβραδυνθεί. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε Χρυσοχοίδη, η συζήτηση περί επιμερισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώνεται η διαδικασία ασύλου και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην αυτών των κρατών πρώτη γραμμή όπως η Ελλάδα, κρύβει την ουσία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη με την ενίσχυση και γενίκευση των απελάσεων που έβηχα αποκαλούνται επιστροφέ, με τη θεώρηση κρατών όπω η Τουρκία, ακόμα και περιοχών στη Συρία ω ασφαλεί τρίτε χώρε ή ασφαλεί περιοχέ, καθώ και με το δραστικό περιορισμό τη ίδια έννοια του πρόσφυγα, αυτό που βασικά θα διαμοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη είναι τι αποφάσει απέλαση χιλιάδων ετούντων άσυλο. Άλλωστε και η δική σα κυβέρνηση έχει ήδη θέσει αριθμητικό στόχο 10.000 απελάσεων έως το 2020 με την παράλληλη ενίσχυση των κλειστών κέντρων. Πώς λοιπόν τοποθετήσετε το γεγονός ότι ο νέος νόμος της κυβέρνησής σας κινείται ακριβώς σε αυτούς τους αντιδραστικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποτελεί εξαίρεση παρανυχίδα, αλλά την ίδια την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προθώντας τον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες, ο οποίος γενικεύεται σε όλη τη χώρα, την καταστολή και με στρατιωτικές δυνάμεις, τις απελάσεις με το δραστικό περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών, ακόμα και με τιμωρητικές διατάξεις, που όλα αυτά αποτελούν βούτυρο στο ψωμί και του εθνικισμού και του ρατσισμού. Ε, Ευχαριστώ πολύ, και από μένα ε, όλη η επιτροπή μας εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζει ότι η ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής έχει αναλάβει πολύ μεγάλο μέρος και βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος όπως γνωρίζει ότι έχει δείξει και έναν ανθρωπισμό για τον οποίο δεν υπάρχει κανένας αντίλογος μας ενημερώσατε ότι εκπονήσατε ένα νέο νόμο για την επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου και προσωπικά οφείλω να βεβαιώσω την επιτροπή ως δικηγόρος μάχημη επί τρεις δεκαετίες ότι αυτός ο νόμος πρωτίστως και κυρίως θωρακίζει και σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων. θέλω να μας πείτε κύριε υπουργέ αν τέτοια νομοθεσία υπάρχει και σε άλλα κράτη μέλη και αν πιστεύετε ότι το γεγονός ότι εδώ και τέσσερα χρόνια με βάση τη δήλωση ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έγιναν μόνο 1.800 επιστροφές. Αν με την δική σας πολιτική της νέας κυβέρνησης θα υπάρξουν περισσότερες επιστροφές ούτως ώστε να τύχει καλύτερης διαχείρισης στο θέμα και επίσης αν πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί και η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ούτως ώστε να μπορούμε να επιστρέφουμε αυτούς που δεν δικαιούνται ασύλου και από την ενδοχώρα, κάτι το οποίο συζητούμε και από τον Αντιπρόεδρο κύριο Μαργαρίτη τη σκηνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, είναι πλέον ξεκάθαρο ποια ήταν τα όρια της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τα όρια ήταν ο, γεωπολιτικό ο γεωπολιτικός εκβιασμός του Ερντογάν στην νοτιοανατολική... Μεσόγειο και Συρία. Από την πλευρά της κυβέρνησης όμως, της ελληνικής κυβέρνησης, θετικό η αποσυμφόρηση των νησιών, άρα ο μη εγκλωβισμός πια προσφύγων όπως η δήλωση αυτή ε, δημιουργούσε ως καθεστώς στην Ελλάδα. Θετικό ότι πάτε να μειώσετε τη γραφειοκρατία στην απονομή ασύλου. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Με εσωτερικό relocation, με εσωτερική μετεγκατάσταση μπορεί η Ελλάδα μόνη της να αντιμετωπίσει ακόμη και την, με την επιτάχυση του, του ασύλου το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης δεν μπορούμε μόνοι μα. Θα υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις το πρόβλημα θα είναι μη διαχειρίσιμο. Σας ζητώ λοιπόν να μα πείτε τι πρωτοβουλίε έχετε πάρει και ζητώ και από του συναδέλφου μου προς τις κυβερνήσεις σας. Πιέστε να υπάρχει επιτέλου ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την κατάσταση. Και δεύτερο ερώτημα. Στα τακτικά κονδύλια υπάρχει χαμηλή απορροφητικότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από τα 613 εκατομμύρια 14-20 έχουν απορροφηθεί 228 εκατομμύρια. Τι προτίθεστε να κάνουμε ως χώρα για να έχουμε αυξημένη απορροφητικότητα και στα τακτικά κονδύλια. Να έχετε υπόψη, παρακαλώ, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Υπουργό και τώρα το να πρέπει να ασχοληθούμε και με το χρονοδιάγραμμα είναι υπερβολή, νομίζω. Σας παρακαλώ, τηρήστε το ένα λεπτό. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Η κατάσταση που περιγράψατε πραγματικά είναι φρικτή και σίγουρα είναι πολύ πιο σοβαρή όταν μιλάμε για τις 34.000 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ΚΙΤ, στα νησιά. Καθημερινά έχω επικαιροποιήσει από κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επιχειρούν επιτόπου στη Μόρια, στη Σάμο, όπως ε, το χάρη, μία μικιό μου γράφει ότι μετά από τη φωτιά στο χώτο του Τσαμός στις 14 Οκτωβρίου πολύ λίγοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν ε, στην υπηρετική Ελλάδα και πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι σήμερα δεν έχουν επίτροπο που να εγγυηθεί την προστασία τους που να μπορεί να τους βοηθήσει νομικά ή να προωθήσει τα αιτήματά τους για επανένωση, για οικογενειακή επανένωση. Επίσης, αυξήθηκαν οι βιασμοί και η άσκηση βίας και υπάρχει και μόνο ένας γιατρός για όλο τον πληθυσμό του ΚΙΤ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς θα προσπαθήσετε να λύσετε την κατάσταση και στο Συμβούλιο για να πεμπλοκάρετε τη συζήτηση για την μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζω κάτι πρωτόγνωρο, ειλικρινά. Έρχεται ο υπουργό μια χώρα που δέχεται το μεγαλύτερο βάρο του προσφυγικού, μα λέει ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό και μη διαχειρίσιμο και το βάζουμε στη γωνιά και το ρωτούμε τι κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνετε γι' αυτό. Γιατί δεν ρωτάμε του εαυτού μα. Γιατί δεν ρωτάμε τι κυβερνήσει τη δικέ μα. Είναι μόνο θέμα τη Ελλάδα. Αυτό καταλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Now, Mr. Ευχαριστώ, κύριο Κώστερ. Δεν νομίζω ότι είναι ελληνικό το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ευρώπη πραγματικά τους απογοητεύει όλους καθώς αποτυχαίνει να δείξει αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και το να βρει μια λύση που να λειτουργεί. Είναι πραγματικά σοκαριστική η κατάσταση και εκπρόσωπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μας ε, έδωσε λεπτομερείς περιγραφές. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε καταπηγόντως δράση. Ακούσαμε τι συμβαίνει με τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τι άλλο κάνετε πέρα από το να στέλνετε όμως επιστολές ε, στους ομολόγους σας. Είμαι απογοητευμένος ε, φυσικά από την έλλειψη αντίδρασης από το δικό μας ε, Υπουργείο Εσωτερικών. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για τις έγκυες γυναίκες, για τους αρρώστους, για τα παιδιά. Είναι καταστροφική και σοκαριστική η κατάσταση. Ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι, να βοηθήσει. Κάτι άλλο που είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι δεν ε, υπάρχουν ε, αντιδράσεις και στο, νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση ότι περιορίζονται γεωγραφικά κάποιοι άνθρωποι. Επίσης ε, και εσείς έχετε κάποια ευθύνη και πρέπει να αναλάβετε δράση εδώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εγώ ήμουν στη Σάμο την περασμένη εβδομάδα για να διαπιστώσω την κατάσταση επιτόπου και πήγε η φούσκα των Βρυξελών επί τόπου. Βέβαια, εγώ είχα ένα επικοδομητικό πνεύμα και όμως με συνέλαβαν και με κράτησαν μια ώρα στο αστυνομικό τμήμα ενώ δεν ήμουν ένοχο για τίποτα. Αυτό είναι ο ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο ε, που ε, θα θέλατε να έχουμε. Όμω, ε, είδα αυτοί οι 600.000 άνθρωποι σε ποια κατάσταση ζουν. Έχουμε εκατοντάδες παιδιά και έγκυε γυναίκες, άνθρωποι που περίμεναν περιμένουν μέχρι το 2021 κάποιοι για ένα ραντεβού για να καταθέσουν την αίτηση ασύλου της. Δεν ε, σέβεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο ε, τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Πατιαρμοστία του ΕΕ για τους πρόσφυγες. Και σήμερα το πρωί είπαμε ότι υπάρχει αποτυχία, δεν λειτουργεί η συμφωνία με την Τουρκία, υπάρχει αποτυχία της πολιτικής ε, των hot spot. Η ελληνική εμπειρία μας το δείχνει καλά και υπάρχει και αποτυχία του Δουβλίνου. Εσείς υφίστατε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ο δήμαρχος ε, της ΣΑΜΟΥ είναι σε απελπισία, καταραίει η οικονομία του νησιού και υπεύθυνη είναι η Ευρώπη. Έτσι λοιπόν εσείς θα απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και ποιες λύσει έχετε σκεφτεί για να βγείτε από το διέξοδο. Κυρία Φόξ, για ένα λεπτό. καλέσατε για αλληλεγγύη και να ασκήσουμε πίεση στι κυβερνήσει σα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λένε ε, μην ανησυχείτε. Ε, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνη, τη μετακυλούμε στον Ερντογάν. Έτσι λοιπόν είναι κατά τη ιδέα ότι μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στα δικά μα εθνικά κράτη, γιατί δεν επιτρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη τέτοιε αποφάσει. Και φυσικά όταν μιλάμε για τον Ερντογάν από όλου του ανθρώπου, τώρα του δώσαμε την εξουσία ότι τα χρήματα εξαγοράζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει και εισβάλλει και σε μια περιοχή στη Συρία και δημιουργεί μια νέα μεταναστευτική πολιτική. Και μετά μπορεί να αναρωτηθούμε γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από την Τουρκία για να έρθουν στα ελληνικά νησιά η κατάσταση στους καταβλισμούς στην Τουρκία πώς είναι. Ίσως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να εντάξει τους μετανάστες ε, στην τουρκική κοινωνία είναι σωστή. Ποιος θέλει να ενταχθεί στην τουρκική κοινωνία που φυλακίζει τους ακαδημαϊκούς, ε, δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου και πρόκειται για ένα αυταρχικό καθεστώς. Νομίζω ότι κάθε μέρος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθά την Ελλάδα και δημιουργεί ένα πρόβλημα που πρέπει όλοι να διαχειριστούμε και θέλω να σας εκφράσω την ελληνική μου. Κύριε Ουρμπάν, να είστε σύντομο για να μπορεί να απαντήσει και ο κύριο Υπουργό, αν και έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν είναι ένα θέμα κλιματικό ούτε τέτοιο είδους καταστροφή. Αποτελεί παροϊόν των πολιτικών αποφάσεων. Τώρα έχουμε 14.000 ανθρώπους στη Μόρια. Αποτελεί προϊόν πολιτικής απόφασης να μην μεταφερθούν σε καταβλισμούς όπου θα ε, έχουν περισσότερη ασφάλεια. Το να ε, αφαιρείτε την ε, πρόσβαση στο ΑΜΚΑ είναι πολιτική της δική σας κυβέρνησης. Μιλώ για τους ασυνόδευτους ελληνίκους δεν μπορούν να εμβολιαστούν με αυτόν τον τρόπο αν δεν έχουν κάρτα υγεία ούτε μπορούν να πάνε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και αυτή είναι πολιτική απόφαση κύριε Υπουργέ εδώ είναι το πρόβλημα ότι λαμβάνετε λανθασμένε πολιτικέ αποφάσει. αν θέλουμε να υπερσπίσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων Α λάβουμε πολιτικέ αποφάσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σύμφωνα με τα δικαιώματα των πολιτών Όπω είπα τώρα έχετε αρκετά προβλήματα αλλά πρέπει να απαντήσετε μέσα σε 10 λεπτά Θα καθυστερήσουμε κάπως για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ, βάλτε τα δυνατά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για τις ε, αγωνιώδεις ε, τοποθετήσεις που κάνατε ε, ρωτώντας και εκφράζοντας την αγωνία σας για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα στα νησιά. Σας ευχαριστώ και για την κριτική που κάνατε αλλά θα παρακαλέσω πολύ η κριτική πάντα πρέπει να έχει μια βάση. Άκουσα τελευταία ε, μια κριτική για το ΆΜΚΑ. Για... Αυτή τη στιγμή λοιπόν στα νησιά, στη Λέσβο και στη Σάμμο εμβολιάζονται όλα τα παιδιά. Πού αφαιρέθηκε η δυνατότητα πρόσβασης υγείας. Αυτό δεν είναι αλήθεια λοιπόν. Όπως δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγεία. Όλοι οι ετούντες άσυλο στη χώρα όλοι οι αιτούντες άσυλο, αυτοί που επίσης έχουν, έχει τελειώσει η διαδικασία τους και αυτόν οι οποίοι έχει τελειώσει η διαδικασία τους και δεν έχουν δικαιωθεί, είναι, έχουν όλοι πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η απάντηση. Όπως επίσης ο νέος νόμος για το δίκαιο του ασύλου προβλέπει υποχρεωτική, υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά των ετούντων άσυλων. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι ε, θα παρακαλέσω πολύ εδώ μέσα να μην αμφισβητεί κανένας και τα δικά μου ανθρωπιστικά αισθήματα που μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από κάποιους εδώ μέσα. Και μάλιστα εγώ καλούμε ως πολιτικός να είμαι και ανθρωπιστής αλλά ταυτόχρονα να είμαι και αποτελεσματικός να είμαι αποτελεσματικό για να υπηρετήσω τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων από τη μια μεριά, την ασφάλεια τη χώρα μου και την ασφάλεια τη Ευρώπη, αλλά και την αξιοπρέπεια τη Ευρώπη, αν θέλετε. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι είσαι ανθρωπιστής και πολύ διαφορετικό όταν επιρρητείς τον ανθρωπισμό και από εκεί κρίνεσαι και κρίνονται και τα έργα σου. Εγώ λοιπόν ως πολιτικός προϊστάμενος αυτού του Υπουργείου θα κρυθώ τελικώς εδώ ενώπιόν σας σε κάποιους μήνες που θα με καλέσει πάλι ο Πρόεδρος από τα έργα μου. Και θέλω να άρω και μια άλλη παρεξήγηση. Ακούστηκε από δύο-τρεις ε, τρία μέλη της Επιτροπής ότι υπήρξε κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ότι ήρθε στο Υπουργείο της Αστυνομίας η αρμοδιότητα της μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό, είναι, αυτό τι είναι εδώ στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια χώρα από εσά, υπάρχει κάποιο Υπουργείο Εσωτερικών του οποίου ηγείται ο Υπουργό τη Αστυνομία, τη Πυροσβεστική, τη Πολιτική Προστασία που δεν είναι ενταγμένη και η μεταναστευτική πολιτική. Μα για όνομα του Θεού τώρα. Τι συζητήσει είναι αυτέ που κάνουμε. Όλα τα Υπουργεία Εσωτερικών έχουν ενταγμένη τη μεταναστευτική πολιτική στι αρμοδιότητέ του. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μια άλλη διευκρίνηση επίση. Ακούστηκε από κάποιο μέλος της Επιτροπής για τα σύνορα. Εγώ δεν αναφέρομαι στα εξωτερικά σύνορα. Δεν αναφέρθηκα στα εξωτερικά σύνορα τα οποία αυτονοήτως πρέπει να ελέγχουμε, να προστατεύουμε ως ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές χώρες και ως Ευρώπη συνολικά. Αλλά αναφέρθηκα στα εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτοί δηλαδή που υψώνουν τύχη σε κάποια χερσαία σύνορα πιστεύοντας ουτοπικά κατά τη γνώμη μου ότι θα μπορέσουν να εμποδίσουν τις ανθρώπινες ροές. Γιατί δεν σταματούνται οι ανθρώπινες ροές και οι άνθρωποι όταν θέλουν να βαδίσουν προς μια κατεύθυνση. Το ζήτημα της Τουρκίας, τρέχω γρήγορα για να προλάβω τα ερωτήματά σας. Το ζήτημα της Τουρκίας και της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιμετωπίζει η ίδια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει στην επικράτειά της περίπου 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Και υποθέτω ότι έχει και άλλους οι οποίοι έρχονται από κάποιες χώρες. Με αυτήν την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για την διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από κυβερνητικές οργανώσεις. Ωστόσο, έχει αναλάβει και μια υποχρέωση να προστατεύει τα σύνορά της. Και αυτό, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι γινόταν μέχρι κάποιο σημείο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ούτε θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που περιγράφω ενώπιόν σας είναι η πραγματικότητα, την οποία πολλοί από εσά έχετε ζήσει. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι η συνέχιση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά με την προϋπόθεση της διασφάλισης των προϋποθέσεων και των συνθήκων που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, αυτή η δήλωση. Δηλαδή η προστασία των συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών των προσφύγων από τη Συρία στο έδαφος της. Έρχομαι πολύ γρήγορα στο ζήτημα, στο ζήτημα του νόμου δύο πράγματα. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι έξι μέρες διαβούλευση, 332 σχόλια εκ των οποίων πρέπει να σας πω σχεδόν τα περισσότερα έγιναν δεκτά. Ορισμένες μάλιστα οργανώσεις και θεσμοί υπέβαλαν προτάσεις και έγιναν από μένα δεκτές όλες οι, οι σημειώσεις που είχαν και οι προτάσεις που είχαν υποβάλει. Και μάλιστα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικώς από δύο κόμματα, από δύο κόμματα καθολικά και από τα υπόλοιπα κόμματα, πολλά από τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν πάρα πολλά άρθρα. Γιατί τι θέλουμε να κάνουμε με αυτόν τον νόμο. Να σας πω τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Για να απαντάμε στην πολιτική πρέπει να απαντάει κανείς με γεγονότα και αποδείξεις και τελικά με αποτέλεσμα. Με στοιχεία λοιπόν του 2019 αυτή τη στιγμή έχουμε 68.000 αιτήσει εκκρεμής. Κάποιος, νομίζω κάποια κυρία Ευρωβουλευτή το είπε, περιμένει τρία χρόνια για να πάρει σειρά για συνέντευξη, για ετών, ετών άσυλο. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μάλιστα με του ρυθμού που υπάρχουν σήμερα, αυτοί οι ρυθμοί οι οποίοι είναι τόσο μεγάλοι που δημιουργούν τα προβλήματα στα νησιά μας. 14.000 προσφυγέ στην αρχή προσφυγών, ο χρόνο σήμερα είναι πάνω από δύο χρόνια και το ερώτημα είναι τι κάνει με αυτού του ανθρώπου όλου. 1.806 επιστροφές σε τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα του νομικού πλαισίου το οποίο ίσχυε μέχρι σήμερα. Και δεν μπορείς, θέλω να το ξανατονίσω αυτό, και επικαλούμε τα ανθρωπιστικά αισθήματα όλων, αλλά ταυτόχρονα και την πολιτική οριμότητα όλων. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλους πληθυσμούς ανθρώπων όταν έρχονται συσσωρευμένοι. Είναι αδύνατο να το κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν δεν τους παρέχεις προστασία. Άρα λοιπόν ως χώρα, ως κράτος δεν μπορείς να τους διασφαλίσεις τα δικαιώματά τους. Και άρα λοιπόν είσαι ελληματικό στην προστασία. Συνεπώς τι πρέπει να κάνεις, να οργανωθείς καλύτερα, να είσαι πιο ταχύς, πιο αποτελεσματικός, να μην στηβάζεις τους ανθρώπους και τελικά να είσαι καλύτερος στην προστασία του ανθρώπου. Θα τελειώσω. έχω ακόμα ένα ζήτημα. Γιατί το βάλατε όλοι. Τι θα κάνουμε με τα νησιά. Υπάρχει ένα σχέδιο. Να μεταφέρουμε τους ανθρώπους από τα νησιά στην ενδοχώρα. Στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ασφαλείς δομές. Σε ξενοδοχεία. Σε διαμερίσματα. Αυτό το εγχείρημα εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος έτσι ώστε όσοι απομείνουν στα νησιά να είναι κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Πρέπει να σας πω ότι η στρατηγική είναι η προτεραιοποίηση και οι πρώτοι που φεύγουν από τα νησιά είναι οι ευάλωτοι, οικογένειε με παιδιά. Οι οικογένειε με παιδιά φεύγουν από τα νησιά για την υπηρετική Ελλάδα. Μέσα από προσπάθεια που γίνεται να δημιουργηθούν δομέ ή να βρεθούν ξενοδοχεία και διαμερίσματα υπάρχει το πρόγραμμα εστία με την υπάτια αρμοστία για 40.000 διαμερίσματα από 1η Πρώτου του 2020, το πρόγραμμα Ήλιος με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για 16.000 σπίτια, δηλαδή εξελίσσεται ένα πρόγραμμα γιατί, κοιτάξτε και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, το μεγάλο ζητούμενο για μας, για την κυβέρνησή μας, είναι το επόμενο βήμα η ένταξη και ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο να μάθουν την ε, ελληνική τα παιδιά αλλά και οι άνθρωποι οι γονείς τους οι οικογένειες να απασχοληθούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τελικά να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας γιατί αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Θα ζήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια και πρέπει να διασφαλίσουμε και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και το σεβασμό στους νόμους, το σύνταγμα της χώρας, το οποίο εφαρμόζουν και σέβονται όλοι οι Έλληνες και τελικά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και πιστεύω πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε θα ξανάρθω υπεύθυνα να καταθέσω το έργο το οποίο θα ξεδιπλώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χρυσοχοίδη. Σας ευχαριστούμε διότι με πάθος αναφερθήκατε στο θέμα. Είναι σαφές ότι έχουμε ένα ανοιχτό θέμα το οποίο δεν είναι ελληνικό για μας, είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Οπότε ο διάλογος επίσης είναι και αυτός ανοιχτός, θα παραμείνει ανοιχτός. Είχαμε διάφορους συνομιλητές που αντιμετώπισαν τη σκληρή κατάσταση υπήρξε σκληρή ανταλλαγή απόψεων, διότι το διακύβευμα είναι πράγματι δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τι θα μας λένε οι Έλληνες Υπουργοί για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Ευχαριστούμε. Και τώρα, χωρίς χρονοτριβή, διότι έχουμε 20 λεπτά καθυστέρηση, πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης. Τέσσερα μέλη του πάνελ θα πάρουν τη θέση τους στο βήμα εδώ θα ξεκινήσουμε παρευθύς. Το τελευταίο σημείο πρωινό θα έχουμε και το απόγευμα συνεδρίαση. Λοιπόν, χαιρετίζουμε τα μέλη του πάνελ. Τρίτο σημείο της σημερινής διάταξης. Ζητώ συγγνώμη από τα τέσσερα μέλη του πάνελ. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Ποια είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά όσον αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκία, Συζητήσαμε ο Γενικό Διευθυντής του Digic Home, η Παρασκευή Μίτσιου, θα μιλήσει, ο Μάικλ Οφλάχερτη, διευθυντή, του ΦΡΑ, η Νίνα Γκρεγόρη, διευθύντρια του Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη Χορηγήσεω Ασύλου, ΕΑΣΟ και Ήρμα Βάσκε τους γιατρούς χωρίς σύνορα εκπροσωπή. Τέσσερα μέλη του πάνελ. Ας ξεκινήσουμε. Αν καταφέρετε 8 λεπτάκια ο καθένας θα μας βοηθούσατε για να μην υπερβούμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας και τις ώρες εργασίας των διαρμηνέων. Ας ξεκινήσουμε. Η κυρία Μίτσιου. Λοιπόν, μπορείτε να ξεκινήσετε παρακαλώ. Καλησπέρα και καλημέρα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι όλες ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Θα είμαι πολύ λακωνικότερη. Πριν έρθω βλέπετε, άκουσα τον Έλληνα Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη που αναφέρθηκε στην κατάσταση. Θα αναφερθώ μόνο στα όσα μας αφορούν. Να πω ότι άκουσα τον Υπουργό που έλεγε ότι είμαστε μόνοι μας. Να πω ότι δεν ήταν μόνη της η Ελλάδα. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στηρίξαμε επιχειρησιακά, οικονομικά την Ελλάδα, άνθρωποι από τη Γενική μου Διεύθυνση, είναι παρόντες, συνάδελφοι από την ΕΑΖΟ, από την Frontex, από την Europol, από τη ΦΡΑΧ, επίση ήταν εκεί. Ίσως όχι μόνιμα η ΦΡΑ εκεί, αλλά η ΕΑΣΟ όμως και η Frontex και η Europol σχεδόν μονίμως εκεί είναι. Τη στηρίξαμε την Ελλάδα οικονομικά επίσης, αλλά η κατάσταση που περιγράφει προηγουμένω βεβαίως δεν είναι βιώσιμη. Ζητήσαμε αύξηση τη της χωρητικότητας στα νησιά, των δυνατοτήτων. Πήγα στα νησιά, το είπα και πριν σε εσάς, σας το είπα όταν η Μόρια είχε 8.500 ανθρώπους πριν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και η κατάσταση ήταν ήδη κρίσιμη τότε, πολύ κρίσιμη. Στη Σάμο ήταν κρίσιμη επί πολλούς μήνες πριν. Τώρα είναι μη βιώσιμη, αναφόρητη. Τι πρέπει να γίνει. Ακούσαμε τον Υπουργό που μίλησε για μεταφορές προς την ενδοχώρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ποιον μετακινούμε στην ενδοχώρα διότι θα σας πω γιατί σε σχέση με τη δήλωση, την κοινή δήλωση στην Τουρκία. Αυτό που αναφέρθηκε ήταν αληθές. Όταν είναι τα οι διαδικασίες, πρέπει να τεθούν προτεραιότητες και πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στη σωστή στέγαση αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί βοηθήσαμε μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ μέσω τη Διεθνού Οργανώσεω Μετανάστε να βοηθήσουμε για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Ήλιο και Εστία και να ετοιμάσουμε πολλού καταβλισμού που χρησιμοποιούνται στην ε, ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα. Τα θέματα υγεία. Ναι, υπήρξαν προβλήματα με τους γιατρούς. Δεν είδαμε όμως κάποιο πρόβλημα ασθενειών πριν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αλλά βέβαια όταν καταφθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, κατάλληλε διαδικασίε, ούτω ώστε αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο να καταχωρηθούν, όχι μόνο να δαχτυλοσκοπηθούν, όχι μόνο να εξεταστούν τα θέματα ασφαλείας, αλλά θέματα υγείας επίσης και υγεία τους. Και πρέπει να φροντίσουμε και τα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα το συζητήσει ο Διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το θέμα των παιδιών περισσότερο την πλευρά μας όμως χρηματοδοτήσαμε και ζητήσαμε την ελληνική κυβέρνηση να γεμίσουν πρώτα τα 2.000 κέντρα στην υπηρετική Ελλάδα να πάνε τα παιδιά, να τους παρασχεθεί η φύλαξη που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργηθεί η στρατηγική για το πώς θα πάνε τα παιδιά. Υπάρχει στρατηγική Παρακολουθούμε στενά τα τεκτενόμενα. Τα παιδιά και τα έχω επισκεφθεί αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά. Τα παιδιά λοιπόν είναι πρόβλημα. 80% παιδιά έχουμε 14 17 ετών παιδιά που φτάνουν. 14 με 17. μετά ενηλικιώνονται. Είναι δύσκολη ηλικία αυτή. Αν δεν μπορούν να δουν ότι έχουν μέλλον τα παιδιά, και το καταλαβαίνει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και εμείς, αν δεν έχουν προοπτικές τα παιδιά, δεν θα βλέπουν μέλλον. Αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνία μας και για τα παιδιά. Και για τη χώρα υποδοχής των παιδιών είναι επικίνδυνο. Εργαζόμαστε εντατικά με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας για τη βελτίωση της κατάστασης. Να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Είναι πολύ κακό να βλέπει κανείς 1600 παιδιά να μένουν σε έναν τόπο που έχει προβλεφθεί για τη στέγαση 300 παιδιών. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Τώρα, οι επιστροφές. συνεργαστήκαμε, εργαστήκαμε πολύ για εθελούσιες επιστροφές. Τι θέλαμε. Να είμαστε σίγουροι ότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας α, λειτουργεί πλήρως. Θέλαμε να έχουμε μετεγκατάσταση, το πετύχαμε. Πάνω από 25.000 μετεγκαταστάσεις είχαμε μετά την έναρξη ισχύω της κοινή δηλώσης Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκία. Βάσει αυτή τη δηλώσεω, θέλαν περισσότερες επιστροφές, αλλά είναι ε, μακράς διαρκεία οι διαδικασίες και είναι άκαμπτο το σύστημα, δίσκαμπτο το σύστημα που ίσχυε και ακόμα ισχύει νομίζω στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Αν ρωτήσω τους Ολλανδούς, όπως έκανα, πόσο χρόνο χρειάζονται οι Ολλανδοί να ολοκληρώσουν μια διαδικασία τέτοια για κάθε άτομο. Μου είπαν αυτοί Τρεις μήνες λίγο πολύ, στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν Πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, καλύτερη χρονική περίοδο από δύο ή τρία χρόνια. Ζητήσαμε τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την νομοθεσία τους, να τη βελτιώσουν, να έχουν καλύτερες διαδικασίες, να γίνεται αξιολόγηση των υποθέσεων αναπερίπτωση αλλά σε ένα εύρυθμα λειτουργούν σύστημα. Και πάνω σε αυτό εργαστήκαμε με, την, ε, με τον Φορέα Προστασία των Μεταναστών για τι επιστροφέ. Πάμε τώρα στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Είπε ο Υπουργό ότι υπάρχει αυτή η δήλωση. Με πολλέ διατάξει και προβλέψει. Και ότι η Τουρκία την εφάρμοζε πριν το καλοκαίρι να σας πω. Εάν έχεις 80-85 από το καλοκαίρι, είναι ήδη αρκετό. Ξέρετε πόσους έλαβε, δέχτηκε η Τουρκία πέρσι, ως πρόσφυγες. Πόσους έλαβε, πόσοι κατέστησαν στην Τουρκία. 300.000. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, μαζί με τη Frontex, και συλλαμβάνουν περίπου 4.000 διακινητές που θέλουν να μετακινήσουν ανθρώπους από την Τουρκία στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Το σύστημα λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο πριν το καλοκαίρι, εξακολουθεί να λειτουργεί. Λοιπόν, πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με τον... Πήγαμε την με τον κύριο Ζιχόφερ και τον κύριο Αβραμόπουλο συνεργαζόμαστε για να μπορέσει να λειτουργήσει στο βέλτιστο δυνατό βαθμό αυτή η κοινή δήλωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πω τώρα. Ελπίζω 1η Δεκεμβρίου να έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι δεν είναι εύκολο για μένα να συνεργάζομαι με δύο ε, επιτρόπους, απερχόμενο και επερχόμενο και σε δύσκολο τομέα. Ελπίζω και με όλους συνεργάζομαι και εργάζομαι σκληρά και με την ίδια την πρόεδρο, την α πρόεδρο, να επιφέρουμε τις αλλαγές που θέλουμε στο μέλλον, να χρησιμοποιήσουμε όλο το καλό προηγούμενο έργο που έχει επιτελεστεί εδώ στο Κοινοβούλιο και είναι πολλή δουλειά που έγινε εδώ. Είναι ένα πρόβλημα, δύσκολο θέμα, δύσκολη κουβέντα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, αλλά πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Now... Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιχού. Κύριο Φλάχερτη, αν τα καταφέρετε σε 8 λεπτά, θα σας ευγνωμονούμε. Βάλτε τα δυνατά σας για να ακούσουμε και τους συντονιστέ, αλλά και τους βουλευτές στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για την πρόσκληση. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη. Θα πρέπει να φύγω μετά την παρέμβασή μου, γιατί έχω να προλάβω ένα αεροπλάνο. Αλλά ο συνάδελφο που είναι εδώ θα μπορέσει να απαντήσει στι ερωτήσει που αφορούν τον οργανισμό μα. Ε, χαίρομαι που τοποθετήσετε αυτή τη συζήτηση για σήμερα. Ξέρετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και ο οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, τα θέματα από το 2016 και έχουμε τώρα ε, μία μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Επισκεπτόμαστε τεχνικά τα κέντρα υποδοχής στα νησιά και εγώ πήγα εκεί πριν 10 ημέρες. Κυρίως ε, προσφέρουμε υποστήριξη στην Ελλάδα ως κράτος μέλος αλλά και στην Κομισιόν και στις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Επιτόπου όπως παραδείγματος χάρη το ΕΑΣΟ και Frontex προσφέρουμε υποστήριξη μέσω παροχής συμβουλών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τεχνική βοήθεια, όπως ε, κατάρτιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ανάλυση της ευαλωτότητας. Επίσης ε, και μέσω παρουσίασης εκθέσεων ε, για την κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη και μέσω επίσημων γνωμοδοτήσεων σε εσά και έχουμε τα λεγόμενα hot spot ε, το 2016, το οποίο υποβάλαμε έκθεση, αλλά και πριν λίγους μήνες επίσης. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τη συζήτηση. Θα αναφέρω κάποια βασικά σημεία σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό. Καταρχήν, 10 μέρες πριν στη Μόρια είχαμε 13.000 ανθρώπους, ενώ έχει σχεδιαστεί η εγκατάσταση για 3.000 και έχουμε 30.000 μετανάστες στα ελληνικά νησιά σε κέντρα που χωρούν 5.000. Ακούσατε την κατάρρευση των βασικών υπηρεσιών. Ο διοικητή ενό καταβλισμού μου είπε ότι η μόνη υπηρεσία που μπορώ να δώσω είναι τρόφιμα και ούτε αυτό το κάνω πολύ καλά. Το θέμα της ε, υγείας αναφέρθηκε, της περίθαλψης. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών, όμως και πάλι δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Έχουμε 10.000 ανθρώπους που περιμένουν ε, έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο. Αναφερθήκε κάποιος ε, στην έλλειψη νόσου, όμως γι' αυτό γίνεται ο πρώτος έλεγχος, για να μην υπάρχει νόσος στους καταβλισμούς. Επίσης υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, ε, το πώς αυτό οδηγεί ε, στην διάχυση των ανθρώπων. Ε, ουσιαστικά έχουμε κάποιες αυτοσχέδιες σχηνές που στείνονται έξω από το χώρο των ίδιων των ΚΙΤ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εγκαταστάσεις υγειονομικές εκεί που στείλουν οι άνθρωποι αυτές τις αυτοσχέδιες σκηνές. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι είναι διευρυμένοι παραμονή. Αρχικά τα hot spot ε, είχαν σχεδιαστεί για να περιμένουν, να οι άνθρωποι για λίγες ημέρες, ε, όχι για να στεγάσουν τους ανθρώπους για πολλούς ε, μήνες όπως συμβαίνει σήμερα. Πράγματι, η κατάσταση των παιδιών τώρα ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που έχουμε στα ελληνικά νησιά, στα ΚΙΤ, είναι η έλλειψη ασφαλών ε, χώρων. Δεν έχουμε αρκετούς ασφαλείς χώρους. Όταν ε, ήμουν πριν 10 μέρες στη Μόρια, είχαμε 10, ε, συγγνώμη, 1000 ε, συνόδευτα παιδιά, όμως υπήρχε χώρος μόνο για 300 παιδιά σε αυτούς τους ασφαλείς χώρους. Δηλαδή, τα 700 παιδιά εκτίθενται σε κάθε είδους κινδύνους. Ε, ένα, μια άλλη διάσταση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που μας ανησυχεί ε, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα του προσωπικού. Δεν αναφέρθηκαν σήμερα, αλλά είναι ήρωες οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις και έχουν πολύ μεγάλο άγχος. Και αυτοί θα πρέπει να προστατευτούν σε αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη στην οποία βρίσκονται. Και επίσης, ως τελευταία κατηγορία θα ανέφερα ε, το θέμα του πληθυσμού των νησιών. Είναι μη βιώσιμη η κατάσταση σε νησιά όπως η Λέσβος, ε, και πραγματικά αυτό προκαλεί ταραχέ και στην ε, τόπια οικονομία. Δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η διάσταση αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, ο Οργανισμός των Μελλοντών Δικαιωμάτων θα προτείνει η δράση για εκτό συγκεκριμένα σημεία αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, πιστεύουμε ακόμη ότι η έννοια του hot spot εξεκολουθεί να έχει νόημα αν λειτουργήσει όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά παραμένει καλή ιδέα, δηλαδή ε, μία και μόνη εγκατάσταση όπου θα γίνονται όλες οι διατυπώσεις κατά την άφηξη. Αλλά για να λειτουργήσει θα πρέπει ε, ουσιαστικά ναι, να διεκπεραιώνει ε, γρήγορα ε, τις διαδικασίες ε, και να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε επίγουσα διαδικασία από αποσυμπίεσης ε, της κατάστασης, ε, μείωση του πληθυσμού και τώρα είναι καλές οι προσπάθειες που γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχουν επίγοντα μέτρα προστασία εντό ε, των ΚΙΤ. Το πρώτο θέμα είναι η παροχή βασικών υπηρεσιών, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης ή, το χάρη, αν υπάρχει έλλειψη σε υποδομές υγιεινής. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα αν δεν αντιμετωπιστούν. Ένα Βασικό μέτρο που χρειάζεται τώρα είναι να έχουμε μεγαλύτερους ασφαλείς χώρους ε, προκειμένου ε, να μπορούν να καλύπτονται όλα τα συνόδευτα παιδιά. Κατόπιν έχουμε μία ομάδα ανθρώπων ε, που ουσιαστικά δεν τη χάνουν καμίας προσοχής και αυτό είναι οι νέοι άνδρες. Και αυτό μας ανησυχεί. Όταν επισκεφτείτε τα κοίτα όλοι θα σας πούν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, της γυναίκες, αλλά κανένα δεν ενδιαφέρεται για τους νεαρούς άνδρες. Και αυτή είναι πραγματική ανησυχία και θα σας ε, εκπλήξει όσοι δεν έχετε επισκεφτεί αυτά τα κίτ ε, πώς χιλιάδες νέοι άνδρες ε, ουσιαστικά βρίσκονται εκεί και δεν έχουν τίποτα να κάνουν και ουσιαστικά αυτό τροφοδοτεί διάφορα περιστατικά βίας που ακούσαμε νωρίτερα. Το επόμενο υπαριθμόν 6 νομίζω είναι, είναι η ανάγκη να κάνουμε καλύτερη δουλειά ε, για να συνεργαστούμε με τον τόπιο πληθυσμό στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ε, των ΚΙΤ. Ε, ουσιαστικά ξέρουμε ότι όταν εμπλέκονται οι τοπικές κοινότητες στη λήψη αποφάσεων λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα. Κατόπιν χρειαζόμαστε να δοθεί προσοχή στις ψυχολογικές ανάγκες του προσωπικού των ε, κέντρων υποδοχής και κατάστασης μας λένε ότι έχουν ε, ε, διαταραχές άγχους αλλά και ότι δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Και προτελευταίο σημείο, πρέπει υπό την επιφύλαξη της συζήτηση για το νέο νόμο ασύλου χρειαζόμαστε πιο ταχείς και δίκαιες διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα. Φρά τον Ιούλιο έδωσε ένα σχέδιο στην κυβέρνηση με 10 σημεία για το πώς θα μπορούσε να θεσπίσει ε, μια διαδικασία πιο ταχεία ε, και δίκαιη, δηλαδή από το πώς μπορείς να έχεις ταχύτερες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων μέχρι να ε, υλοποιήσεις ταχύτερα τη διαδικασία και να έχεις, παραδείγματος χάρη, και καλύτερη κατάρτιση και προβλεψιμότητα των δικασιών για τα παιδιά, συγκεκριμένα ζητήματα. Καταρχήν υπάρχει ένας νέος νόμος επιτροπίας ε, που ε, ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο οργανισμός έδωσε ε, συμβουλές, είναι καλός νόμος, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή και νομίζω ότι πρέπει σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή, γιατί αυτό θα δημιουργήσει και τις συνθήκε για να βγουν τα παιδιά από αυτά τα κέντρα και να πάνε σε ασφαλείς χώρους. Και τέλος, ό,τι αφορά τα παιδιά, Ήδη ακούσαμε τον Υπουργό σήμερα το πρωί για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ζητήσει από όλα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν κάποιους ασυνόδευτους ενηλίκους. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετική ιδέα, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Σίγουρα δεν θα λύσει το ευρύτερο πρόβλημα, αλλά είναι ένα σημαντικό σημείο εισόδου για τους πλέον ευάλωτους και καθώς ε, ξέρετε ότι το πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά. Θα κλείσω εδώ, Πρόεδρε. Απλώ να πω και αυτό είναι προσωπικό σχόλιο, δεν εκπροσωπώ τον οργανισμό εδώ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η κατάσταση των μεταναστών σε ελληνικά νησιά αυτή τη στιγμή είναι ε, ε, το πιο ανησυχητικό θέμα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουμε οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική η δήλωση που κάνατε. Θα περάσουμε τώρα στην Ινά Γκρεγόρη, εκτελεστική διευθύντρια της ΕΑΣΟ. Επειδή οι διερμηνείς θα σταματήσουν στις 12.30, θα ήθελα να σας ζητήσω, μια που θα έχουμε και απογευματινή συνεδρίαση, να είστε σύντομοι. Μετά τις 12.30 θα συνεχιστεί η συνεδρία στα αγγλικά. Κύριε Γκρεγόρη, σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Μιλώ γρήγορα εξάλλου, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Είχα ήδη την τιμή να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ κατά την παρουσίαση ε, της ε, δουλειάς της ΕΑΣΟ και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε ξανά για να τοποθετηθώ για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην Ελλάδα. Η ΕΑΣΟ έχει βελτιώσει την επιχειρησιακή υποστήριξη στην Ελλάδα από το 2011, αλλά το 2015 αύξησε την ε, βοήθεια. Εκείνη την εποχή ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, από την ε, ΕΑΣΟ να βοηθήσει στον, στην επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα hotspot. Έπειτα, μετά την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ο αριθμός των εισερχομένων μειώθηκε, όμως παραμένουν οι μεγάλος και η Ελλάδα, όπως ακούσαμε πολλές φορές, χρειάζεται στήριξη τα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερα τους ε, καλοκαιρινούς μήνες αυξήθηκε η ε, πίεση για την αύξηση συγχωρητικότητας και για την γρήγορη επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Γι' αυτό και η ΕΑΣΟ συνεχίζει να στηρίζει την Ελλάδα και ελπίζω αυτή η αυξημένη στήριξη να συνεχιστεί και το 2020. Οι επιχειρήσεις της ΕΑΣΟ στην Ελλάδα είναι, καλύπτουν ένα εύρος τομέων. Στηρίζουμε τις ελληνικές αρχές στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο της ε, αίτηση ασύλου, αλλά και σε θέματα υποδοχής. Ε, βέβαια, στα θέματα υποδοχής έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Περίπου 500 εργαζόμενοι της ΕΑΣΟ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, παρέχουν καθημερινή στήριξη σε 36 σημεία σε όλη την Ελλάδα από τους 500 ε, ε, εργαζόμενους υπάρχουν και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη, υπάρχουν ε, συμβασιούχοι, υπάρχουν διερμηνείς, αλλά και μόνιμοι υπάλληλοι σε αυτά τα 36 σημεία της χώρας. Να αναφέρω εδώ ότι ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιεί η ΆΣΟ για να Εργαστή στην ε, Ελλάδα είναι χαμηλός. Έχει παρατηρηθεί μία μείωση εδώ και αρκετά χρόνια και τώρα έχουμε μία μείωση της τάξης του 13%. Δηλαδή, μόνο το 13% των ε, εργαζόμενων της ε, ΕΑΣΟ προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο δισταγμός. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θέλω ούτε να κάνω εικασίες για την αλληλεγγύη των εκατών μελών, όμως η ΆΣΟ έχει ως καθήκον να παρέχει ε, επιχειρησιακή στήριξη. Τι κάνουμε τώρα στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, Παρέχουμε τη στήριξη στις ελληνικές αρχές για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, πρωτοβάθμια και στα σύνορα δηλαδή, αλλά και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας. Ε, έχουμε στόχο να αποφορτίσουμε τις ε, αρχές και να εφαρμόσουμε το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή, με την παροχή πληροφοριών, με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για χορήγηση ασύλου και με την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων. Το 2019 έχουν καταγραφεί πάνω από 30.000 αιτήσει από τους υπαλλήλους μας, πάνω από 6.000 συνεντεύξεις έχουν γίνει και πάνω από 1.500 καταληκτικά σχόλια, απορίσματα έχουν ε, εκπονηθεί από εμάς. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση ασύλου βέβαια παραμένει ε, απόφαση των ελληνικών αρχών. Δεν θέλουμε λοιπόν να παρέμβουμε στις ε, εθνικές αρμοδιότητες στο θέμα αυτό. Επίσης, στηρίζουμε την ε, μονάδα Δουβλίνου στην Αθήνα, προσπαθούμε να, ώστε να εφαρμόζεται ο κανονισμός και επεξεργαζόμαστε πολλές αιτήσει. Η ΕΑΣΟ επίσης παρέχει στήριξη στις ε, αρχές σε περιπτώσεις ε, προσφυγής. Παρέχουμε νομική κατάρτιση. Έχουμε καταρτήσει πάνω από 300 φακέλους ε, περιπτώσεων έφεσης στη διαδικασία σύλλου. Όπως σας είπα, έχουμε περιαρισμένες δυνατότητες και προσπαθούμε μέσω πιλωτικών προγραμμάτων να στηρίξουμε τις αρχές και στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη ΣΑΜΟ. Επίσης, παρέχουμε στήριξη στις ε, εγκαταστάσεις υποδοχής, στις πιο ευάλωτες ομάδες, τους ασυνόδευτους ανήλικους, τα παιδιά και ε, λειτουργούμε ως διεύλωση επικοινωνίας μεταξύ των ε, hotspots, Φυσικά, οι προκλήσεις είναι υπαρκτές και επιμένουν. Ε, ο Υπουργός σας εξήγησε την ε, δική του οπτική γωνία. Από τη δική μας πλευρά, στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε μία ασφαλή και ταχεία διαδικασία ασύλου. Βέβαια, η ΆΣΟ χρειάζεται στήριξη και όπως σας είπα υπάρχει έλλειψη προσωπικού από τα κράτη-μέλη, το οποίο πρέπει να αλλάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στα hot spot. Το θέμα αυτό παραμένει μια πρόκληση. Υπάρχουν εντάσεις που δημιουργούνται ιδιαίτερα εξαιτία τη μεγάλη αναμονή για την επεξεργασία μιας αίτηση ασύλου και φυσικά εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ πολύ σύντομα στο ε, σχέδιο κανονισμού για το άσυλο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δραστηριοποιούμαστε εντός της εντολής μας και εντός της νομοθεσίας. Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να φτάσει στα χέρια σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκετά σύντομα και ελπίζουμε με τον τρόπο αυτό να βελτιωθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν μέσω μιας ενισχυμένης εντολής και έτσι ίσως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την Frontex το έργο της. διότι υπάρχει μία αλληλεξάρτηση και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα, να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ε, στέγασης της ΕΑΣΟ στην Ελλάδα. Ε, σας ε, πω ότι αυτή η κατάσταση έχει κάποιο καιρό που κρατάει. Οι αρχές η υπηρεσία μας δεν έχει κάποια συγκεκριμένη έδρα ή κάποια γραφεία στην Ελλάδα και εδώ να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές αρχές και τον Υπουργό Χρυσοχοίδη αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Κουμουτσάκο οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ελπίζω οι υπογραφές για την στέγαση να ε, γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Χρειάζεται βέβαια και η ενό σωστού πλαισίου και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη που μας παρέχει, γιατί δίχως αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ε, βρίσκομαι επικεφαλή ΕΑΣΟ, δηλαδή από τον Ιούνιο φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Γκρεγόρη. Η κυρία Βάσκε εκπρόσωπο ε, των γιατρών σύνορα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μας καλέσατε σε αυτή τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ επί πιο συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία. Αυτά που παρατηρούμε με τις ιατρικές ομάδες επιτόπου. Ξεκινήσω με μια δήλωση ανθρωπιστικού είδους είναι μια τραγωδία, έχω να πω, ανθρωπιστικά η κατάσταση. Πρέπει ε, να, αν το έχουμε αποτροπή αντί να έχουμε σωστές συνθήκες υποδοχής, έχει συνέπειες για τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα ελληνικά νησιά. Οι ιατρικές ομάδες των γιατρών χωρίς σύνορα στη Λέσβο, στη Σάμο και στη Χίο καθημερινά αντιμετωπίζουν ε, σοβαρότατες υποθέσεις ευαλώτων ανθρώπων και παιδιών και η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Ακούμε τις προσπάθειες αλλά δεν βλέπουμε επιτόπου πραγματικές βελτιώσεις. Να πω ότι η φυσική και η ψυχική υγεία επιδεινούνται λόγω των συνθήκων διαβίωσης. Λόγω της έλλειψης υγιεινής αλλά και λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από το σύστημα της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ενώσης Τουρκίας οι άνθρωποι όλο και περισσότερο ε, είναι σε κατάσταση κράτησης, σε ένα νομικό κενό. Και αυτό επηρεάζει την ψυχική του υγεία, αλλά και τη φυσική του υγεία. Να τονίσω δύο βασικές στοιχές για την υγεία. Το ένα είναι η ψυχική υγεία, κάτι που ήδη αναφέραμε το 2017. Ήδη οι γιατροί στο σύνορα, χωρίς σύνορα αναφερθήκαν στην κρίση όσον αφορά την ψυχική υγεία στα νησιά. Το 2018 ετοιμάσαμε ενημερωτικό έγγραφο όπου εκεί τονίζαμε τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που επηρεαζόταν ή που υπέφεραν από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Το 2019 η κατάσταση είναι χειρότερη. Το τελευταίο εξάμεινο στη Λέσβο 20% των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας. Εντός των ασθενών έχουμε 50% από αυτούς που είναι θύματα βασανιστήριων ή κακομεταχείριση 30% των ασθενών με ψυχικά προβλήματα είναι θύματα σεξουαλική βία στην περίπτωση των παιδιών. Έχουμε πάνω από ένα τέταρτο από τα παιδιά που είναι, έχουν ψυχική ασθένεια που έχουν ε, αυλάπτουν τον εαυτό τους. Κάποια από αυτά προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν και κάποια ήταν μικρότερα από 10 ετών. Ε, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στα ελληνικά νησιά. Ήδη αναφέρθηκε η κατάσταση των παιδιών και πράγματι προβληματιζόμαστε όσον αφορά την υγεία και την προστασία των παιδιών. Να υπενθυμίσουμε ότι 50% των ανθρώπων που είναι παγιδευμένα στα νησιά είναι παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη στο... σε αυτά πρέπει να γίνουν. Ιατρικά στοιχεία. Ένα τρίτο από τα παιδιά ζουν σε κατασκηνώσεις ε, και κατασκευάσματα με πλαστικό στα νησιά. Αναφερθήκαμε ήδη, αναφέρθηκαν τα προβλήματα με τον επιπληθισμό στα κέντρα υποδοχής. Ε, μια τουαλέτα για 300 παιδιά στη Σάμο μια τουαλέτα για 200 άτομα σε κάποιες περιοχές ε, στη Λέζο και τα πρότυπα είναι 20 άτομα ανά τουαλέτα. Και έτσι ασθενούν τα παιδιά υπό αυτές τις συνθήκες. Και συγκεκριμένο πρόβλημα ε, παιδιά με περίπλοκα ιατρικά προβλήματα που δεν έχουν επαρκή θεραπεία στα νησιά και θα πρέπει να παραπεμφθούν. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα να παραπεμφθούν στην κατάλληλη θεραπεία. Και ενήλικες αλλά και παιδιά δεν μπορούν να δεχτούν την κατάλληλη θεραπεία. Κάτι που ανέφερε και ο Υπουργό να αναφέρω κι εγώ. Σήμερα, ακόμα σήμερα, η πρόσβαση στην περίθαλψη για τους μετανάστες στα ελληνικά νησιά βασίζεται πολύ σε οργα... εθελοντικές οργανώσεις με πολύ λίγα μέσα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ακόμα βασίζομαστε σε εθελοντικέ οργανώσει για την περίθαλψη. Κάτι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό. Και άλλο σημαντικό σημείο να τονίσω όλο και περισσότεροι άνθρωποι παγιδεύονται στα νησιά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Να χρησιμοποιήσω τα δικά μας θετικά στοιχεία. Σήμερα, πάνω από 45% των ασθενών των γιατρών χωρίς σύνορα στη Λέσβο είναι πάνω από εξάμεινο στα νησιά και κάποιοι πάνω από 1,5 χρόνο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό επηρεάζει την υγεία τους και την ψυχική τους υγεία. Παγιδεύονται οι άνθρωποι λοιπόν στα νησιά λόγω των προβλημάτων των ασυνεπιών που δημιουργούνται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ενώσεω Τουρκία, από το σύστημα που δημιουργήθηκε από την κοινή δήλωση, που δεν προσαρμόζεται αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα τη μετανάστευση και δεν καλύπτει τι ανάγκε προστασία των ευαλωτών ανθρώπων. Και φοβόμαστε, όπω αναφέρθηκε και πριν, ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω μέσω τη νέα νομοθεσία. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη πτυχή που θα θέλαμε να περιγράψουμε και να τονίσουμε, διότι έχουμε και τις πληροφορίες κατάλληλες, είναι η αξιολόγηση του ευάλωτο, της ευαλωτότητας των ανθρώπων. Παραδείγματο χάρη, μέσω στοιχείων το 2018, 70% των ασθενών με ψυχικά προβλήματα στη Λέσβο δεν είχαν ε, εντοπιστεί, δεν είχαν καταταχθεί σαν ευάλωτα άτομα και φοβούμαστε ότι αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω το πρόβλημα κάποιες ασθένειες δεν εντοπίζονται, δεν υπάρχει κατάλληλη διάγνωση και αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Είχαμε περιπτώσεις σοβαροτάτων ασθενούντων που επεστράφησαν ή απελάθησαν προς την Τουρκία. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τι άλλο να πω. Τέσσερα χρόνια πέρασαν και πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει κάτι να κάνουμε συστάσεις συγκεκριμένες. Να χρησιμοποιήσω διαφορετικούς όρους από ό,τι μέχρι τώρα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει κατεπίγουσα εκένωση των ανθρώπων από τα hot spots. Πρέπει ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη τους ευάλωτους ανθρώπους και τα παιδιά που χρειάζονται κατεπηγόντως ιατρική περίθαλψη, αλλά η εκένωση είναι κάτι ευρύτερο από αυτό. Για μας δεν είναι μόνο η μεταφορά που αναφέρθηκε, δεν αρκεί η μεταφορά προς την ε, υπηρετική Ευρώπη, από τα, νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και εκένωση προς τίτες χώρες και προς την Ευρώπη. Προς άλλες χώρες της Ευρώπης. Μεταεγκατάσταση. Αύξηση του ρυθμού μεταεγκατάσταση προς άλλες χώρες της Ευρώπης. Χρειάζονται και τα δύο. Και κάτι άλλο που χρειάζεται και το επαναλαμβάνουμε σαν ανθρωπιστική οργάνωση είναι να, να σταματήσουν αυτοί οι γεωγραφικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τα κράτη με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις. Εάν δεν σταματήσει αυτό θα συνεχιστούν τα προβλήματα. Αντί να να ισχύει αυτό το ίδιο σύστημα, θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα σύστημα δίκαιο ασύλου, δίκαιο σύστημα ασύλου ευρωπαϊκό που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται και την προστασία τους. Έχουμε ευρύτατη τεκμήριωση. Θέλουμε να γνωστοποιήσουμε την πραγματικότητα στα ελληνικά νησιά. Επανειλημμένα προσπαθήσαμε, ελπίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει αλλαγές. Αλλά με θλίψη μου λέω ότι δεν είδαμε αλλαγές. Ελπίζω να σημειωθούν αλλαγές. Το σύστημα όμως πρέπει να αναθεωρηθεί. Με το παρόν σύστημα όλες οι προσπάθειες θα είναι στήρες, δεν αρκούν, δεν θέμα αριθμών. Είναι κάτι παραπάνω από αριθμούς. Είναι θέμα λογικής. Δηλαδή λέμε κλείνουμε τα σύνορα και διορθώνεται το σύστημα. Ε, εν τω μεταξύ κλεισίματος συνόρων και διόρθωση του συστήματος σημειώνονται θύματα, υπάρχουν θύματα. Και αυτά είναι άνθρωποι, είναι θύματα από πλευράς ανθρωπιστικής. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάσκη. Να περάσουμε τώρα στους συντονιστές. Δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ έχετε το λόγο και μετά θα έχουμε και δυνατότητα για τους υπόλοιπους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Κλείνουμε τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Πέρα από τους συντονιστές έχουμε κύριο και στο Mrs and Mr. το And you're Τέλος. Γιατί διαφορετικά θα είναι αδύνατον να τα καταφέρουμε. Παρακαλώ. Ξεκινήστε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο για αρκετά θέματα. Αλλά καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε σήμερα το πρωί. Θέλω να επικεντρωθώ και σε αυτό που είπε η Γενική Διευθύντρια. Ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πώς εσείς βλέπετε να προχωρήσει το Συμβούλιο για μια σειρά θεμάτων που έχουν μπλοκαριστεί στην τελευταία θητεία. Φυσικά είμαστε σε άτυπες συζητήσεις ε, και με τους ε, απερχόμενους και με τους επερχόμενους επιτρόπους για το τι θα γίνει με τα πακέτα που έχουν μπλοκαριστεί για το αν θα πρέπει να περιμένουμε νέε πρωτοβουλίε και για το αν εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε επισήμω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε εμάς με νέες πρωτοβουλίε. Γιατί ενίοτε φοβάμαι ότι έχουμε πολύ ευαίσθητες πλειοψηφίες ε, σε θέματα οριζόντια και γεωγραφικά και πολιτικά και δεν θέλω να χαθεί αυτό. Και επίσης ε, οι συντονιστές θα θέλαμε να δούμε πού βρίσκεται το κοινό έδαφος και εσείς είστε σε κατάλληλη θέση να επανέλθετε σε εμά και να δούμε αν εξακολουθεί να υπάρχει συμφωνία αυτή που βρέθηκε εδώ και στο Συμβούλιο και να πιέσουμε, γιατί φοβάμαι ότι θα επανερχόμαστε στο Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες, έχουμε βάλει στην κορφή του θεματολογίου το μεταναστευτικό σε όλα τα κρατημέλη και φοβάμαι ότι ε, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσει στη αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι μιλάμε για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά εδώ και πολλή ώρα. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα-δύο θέματα. Η μία ερώτηση είναι τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πρόσφυγες στα νησιά τώρα που έρχεται ο χειμώνα. Ακούσαμε ότι είναι καταστροφική η κατάσταση. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν συγκεκριμένα. Η δεύτερη ερώτηση. Ε, ίσως έχει να κάνει με το υπερβολικό άχθος ε, των αρχών. Έχει αλλάξει εντωμεταξύ μεταξύ η κατάσταση και τώρα μπορεί να γίνει και η καταγραφή και ένα μέρος ε, της αίτηση, της διαδικασίας της υποβολής αίτηση στα νησιά ή χρειάζεται να πάει κάποιος στην Αθήνα για να γίνει αυτό. Γιατί αν αλλάξει αυτό μπορεί να επιταχύνει και τη διαδικασία. Επίσης, θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό η Κομισιόν και το ΕΑΣΟ μπορούν να βοηθήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων στα νησιά και τι μπορούν να κάνουν και τα άλλα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση και να βοηθήσουν την Ελλάδα καταρχήν να υλοποιήσει τη διαδικασία σύλλου αλλά και τις επιστροφές και να τους παρέχουν περισσότερη στήριξη σε ό,τι αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στοντοράκη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα καταρχήν. Ευχαριστώ την Γενική Διευθύντρια και όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Βλέπω ένα κοινό στοιχείο στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Νομίζω κάποιος το είπε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια, αφού ξεκίνησε η κρίση του μεταναστευτικού, ε, έχουμε τις ίδιες ad hoc γρήγορες λύσεις που είχαμε βρει τότε για να επιληθεί η κρίση. Και αναφέρομαι στη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και στο ότι εφαρμόζεται στην Ελλάδα, στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Και φυσικά εδώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων και να προσθέσω τις δύο ερωτήσεις μου. Το ένα έχει να κάνει με το μέλλον. Και τι πιστεύει η Κομισιόν ότι είναι μια βιώσιμη λύση. Ακούσαμε για το σύμφωνο για τη μετανάστευση, ζητήσαμε αν την Επίτροπο να μας αναφέρει το περιεχόμενο για το σύμφωνο δεν έχουμε λάβει πολλές λεπτομέρειες. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε σε διαδικασία κατάρτισης. Όμως θα ήθελα μια πρόβλεψη για το πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα για το να επιτευχθούν αυτές οι βιώσιμες λύσεις που χρειάζεται κατεπηγόντως η Ελλάδα καταρχήν. Και η δεύτερη διάσταση της ερώτησης είναι ότι έχουμε μία νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Σε εσά απευθύνομαι, κυρία Μίχου, λοιπόν πέρα από τις βιώσιμες λύσει που ελπίζουμε να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ εμεί από την πλευρά μας θα βάλουμε τα δυνατά μας για να ελοπιθεί αυτό, πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα. Πώς ε, βλέπετε τις λύσεις που θα πρέπει να θετήσει το ελληνικό σύστημα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με το χρόνο της διαδικασίας κατάθεσης ασύλου, το ότι επαναλαμβάνονται πολλά στάδια της διαδικασίας χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος λόγος. Και πολλές φορές καθυστερούν διαδικασίες ε, τρία χρόνια, περιμένουν άνθρωποι την απόφαση ε, να επιληθεί η καταστασή του ή την επιστροφή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τέσσερις ομιλητές ε, για την επισκόπηση αυτής της φρικτής κατάστασης στα ελληνικά νησιά που υπογραμμίστηκε από πολλούς ομιλητές. Είναι αλήθεια ότι η ε, κατάσταση συγκράτησης ε, και ε, υπερβολική σώρευση ανθρώπων στα ελληνικά νησιά οφείλεται και στο θέμα της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Φοβάμαι όμως τι θα γίνει αν έχουμε και άλλες αφήξεις. Θα υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες για επιστροφές στη Τουρκία. Αν δείτε και τις απειλές απέλασης σε χώρες ασφαλείας, και δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα με την αναχέτηση γιατί τελικά ε, απλώς ε, οι άνθρωποι δεν είναι ασφαλείς ε, και τραυματίζονται. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κοινή ευθύνη. Είναι σοκαριστικό ότι έχουμε μόνο 13 εθνικούς εμπειρογνώμονες στο ΕΑΣΟ και έχουμε μόνο 1.100 περιπτώσεις ε, μετεγκατάστασης το τελευταίο έτος. Πώς μπορούμε λοιπόν να επιταχύνουμε τα μέτρα μετεγκατάστασης ε, στα άλλα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να ε, διορίσουμε περισσότερους εμπειρογνώμονες, εθνικούς εμπειρογνώμονες στο ΕΑΣΟ. Επίσης, αν λειτουργούσε το σύστημα θα είχαμε αυτή την άμεση ανάπτυξη από το ΕΑΣΟ. Θα μπορούσαμε να έχουμε και γιατρούς, νομικούς, διερμηνείς, όλες αυτές οι υπηρεσίες που επιγόντως χρειάζονται στα ελληνικά νησιά θα μπορούσαμε να τις έχουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια διαδικαστικά και δεν υπάρχει έλλειψη όλων αυτών που ανέφερα. Και έχω και μια ερώτηση για την ελληνική νομοθεσία που μόλις υιοθετήθηκε. Πώς ε, οι ομιλητές θεωρούν, πώς βλέπουν να έχει αντίκτυπο αυτή η νομοθεσία θα επιδεινώσει την κατάσταση και πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μια ακόμη ερώτηση, όχι μόνο για το θέμα της μετεγκατάστασης, αλλά και οι διαδικασίες οικογενειακής επανέρωσης είναι πάρα πολύ αργές. Ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια οι οικογένειες. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να πιέσει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή της ομιλήτριας και μπορώ να πω ότι κανένας δεν θα αμφισβητήσει εδώ τον δραματικό χαρακτήρα της κατάστασης που περιγράψατε. Όμως, παρόλε τις προσπάθειες που κάνατε, υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα συνέστημα ότι όσο περισσότερο μέσα ε, ενεργοποιούνται οι πόρτες επιτυχίας των προσφύγων, όλο περισσότεροι πρόσφυγες θα έρχονται. Και τελικά θα παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε χώρα, όπως συμβαίνει τώρα στα ελληνικά νησιά. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μια γενική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε απέναντι στη μετανάστευση, γιατί στην πραγματικότητα και εμείς και οι κυβερνήσεις έχουν μια ανησυχία και θέλουν να προστατεύσουν το δικό τους πληθυσμό. Και όπως ε, είπε στη Γαλλία σοσιαλιστής ε, Πρωθυπουργό, δεν μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τη μιζέρια όλου του κόσμου και τώρα εδώ εσείς προσπαθείτε να διαχειριστείτε αυτό ζητάτε περισσότερα μέσα όσο περισσότερα μέσα έχουμε τόσο περισσότερους ανθρώπους θα έχουμε να διαχειριστούμε και τόσο μεγαλύτερα δράματα θα υπάρχουν και σε σχέση με τους πρόσφυγες και σε σχέση με το προσωπικό και σε σχέση με τους ντόπους πληθυσμούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική πολιτική και να πράξουμε έτσι ώστε να είμαστε ε, πραγματικά αυστηροί στο θέμα της υποδοχής, γιατί ξέρουμε ότι μεταξύ αυτών των προσφανών υπάρχουν ε, και πάρα πολλοί ετούντες άσυλους, που, τον οποίο έτσι θα απορριφθεί και θα είναι άνθρωποι που θα παραμείνουν σε παράνομη κατάσταση και όπως έκανε η ελληνική κυβέρνηση, ε, όλες ε, οι κυβερνήσεις που θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτόματα θα υφετήσουν νομοθεσία όλο ένα και πιο αυστηρή. Ίσως ε, δεν είστε εσείς κατάλληλοι να απαντήσετε σε αυτό, όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική. Το να κάνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα Ελντοράντο, γιατί ε, πρέπει να αποφύγουμε να έρχονται με αυτή την πεποίθηση και τελικά να καταλήγουν σε δράματα ή σε θάνατο. Τελικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της μετανάστευσης και μέσω δράσεων της κυβερνήσεων. Ευχαριστώ κύριο Σερβανίτης για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μίκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ καλή περιγραφή που μας κάνατε. Θέλω να σα πω δύο πράγματα και θέλω να τονίσω και στου συναδέλφου μου εδώ ότι δυστυχώ ο Υπουργό κ. Σαχοϊδής είπε τη μισή αλήθεια σε ό,τι αφορά στον νόμο και θα αναγκαστούμε να κάνουμε τεκμηρίωση προ όλου τους βουλευτές γιατί ο νόμο δεν είναι αυτό που περιέγραψε ο κ. Σαχοϊδής. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο άσυλο όπω τα περιέγραψαν οι συνάδελφοι βουλευτέ από το Ρηνιού, του Πρασίνου και του Σοσιαλιστέ. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχει ένα νέο status quo στη νέα εξουσία στην Ελλάδα. Να κάνουμε στους πρόσφυγες τη ζωή δύσκολη. Ούτε άμκα, ούτε σχολεία, ούτε εκπρόσωπος του ΙΕΣ σε Επιτροπές Ασύλου. Οι εκπρόσωποι σα στην Αθήνα ε, από τους γιατρούς χωρίς σύνορα κατήγγειλαν αυτό τον νόμο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το νέο νομικό πλαίσιο, επιμένω, βοηθάει. Δεύτερο που θέλω να σημειώσω. Η κατάσταση ήταν άσχημη. Μέχρι και το Μάιο. 5.000 άνθρωποι σε δομές στη Μόρια, πήγα στη Μόρια, είδα τι έγινε. Ξέρω τι γίνεται. 5.000 άνθρωποι σε δομές των 3.000. Απαράδεκτο. Ο κύριος Χρυσογοίδης πήγε τον Ιούνιο στη Μόρια σε 7.000 κόσμο και είπε ότι ήταν ικανοποιητικέ συνθήκες. Πήγαμε με τον συνάδελφό μου από τους πριν από ένα μήνα ήταν 14.001. 1.200 συνόδευτα παιδιά. 11 μόνο κοινωνική λειτουργή. Σοβαρά ζητήματα. Σήμερα μαθαίνω ότι είναι 17.000. Αυτή η πολιτική της πολιτική αιμονή τη ε, αποτροπή φαίνεται ότι δεν βγαίνει τελικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, καταγγέλλοντα, δεν σα αφορά τόσο συναδέλφου. Ξέρετε, κάτω στην Ελλάδα, βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία επικροτούν κινήσει γιορτών έξω από τα κάμπ, σφάζοντα και δίνοντα κεφάλια, κεφάλια γουρουνιών για να προκαλέσουν του μουσουλμάνους. Όνομα αυτού κύριο Κυρανάκη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πρόβλημα κάτω πολιτικο πολιτικο-ιδεολογικό πια. Η ερώτησή μου είναι μία. Και επιμένω. Το νέο πολιτικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, σα εξυπηρετεί στη δουλειά σα. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε μαζί σα για να καταθέσει νέο νόμο. Sorry. Okay. Λοιπόν, Αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος ε, γύρος, καλύτερα να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους καλεσμένους να απαντήσουν και σας ενημερώνω ότι μετά τις 12.30 όλα θα γίνονται στα αγγλικά. Παρακαλώ. Πείτε μου, ε, ξέχασα κανέναν. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου του κ. Προκατσίνη, ο οποίο απουσιάζει. Ωραία. Ωραία, θα λάβετε το λόγο λοιπόν εκ μέρου τη ομάδα CCR. Το πολύ δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα αυτά που είπατε και τα εξή συμπεράσματα βγάζω. Εσείς όπως και εγώ έχετε την άποψη ότι η κατάσταση στη... στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαράδεκτη και εγώ στην θέση σας νομίζω το ίδιο θα έκανα. Όμως ε, δεν μπορούμε να του αφήσουμε όλους ανεξέλεκτα. Η Ευρώπη δεν αντέχει αυτή την πίεση. Υπάρχει μια τεράστια έλλειψη στέγασης. Ο αριθμός των αστέγων έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Η αστυνομία ε, δεν προλαβαίνει να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν περιστατικά εγκληματικότητα και μέσα σε αυτούς τους καταβλισμούς. Ακούσαμε και τις αναφορές στο μοντέλο της Αυστραλίας. Βέβαια, νομίζω πως τα πράγματα πρέπει να ε, τα αντιμετωπίσουμε από την αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω από σας πού βρίσκονται τα όρια, τι μπορεί να καταφέρει η Ευρώπη δεδομένου ότι υπάρχουν τόσο πολλοί, πολλοί άνθρωποι στην Μέση Ανατολή και στην ε, Αφρική που έχουν ανάγκη. Θα, αυξηθούν, ε, ε, θα αυξηθεί ο πληθυσμός και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Μωράης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που είπαν οι προσκεκλημένοι αναφέρθηκαν στους ε, πολλούς εργαζόμενους από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η Γενική Διευθύντρια αναφέρθηκε στην ε, κατάσταση, τη χαρακτήρισε ως ε, κρίσιμη ή ως δυσβάσταχτη. Ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτή τη στιγμή βρέχεις πρόθεσμα. Στη Μόρια έχουμε φτάσει σε σημείο έκτακτης ανάγκης είναι πραγματικά μια πληγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που συμβαίνουν εκεί. Διότι είναι ακραία η κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ Γενική Διευθύντρια, είναι το εξή. Όταν γίνεται λόγος για μετεγκατάσταση δεδομένων όσων συμβαίνουν στη Μόρια, ε, πώς είναι η έκβαση αυτών των ε, συζητήσεων. Δεν είναι πάντα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό, ειλικρινά, νομίζω ότι μπορούμε από τη μία να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να δείξουμε συμμόρφωση, αλλά τι ακριβώς έχει υποθεί. γνωρίζουν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εκεί. Στην Ελλάδα, από την άλλη, υπάρχει νέος νόμος και αντικειμενικά μιλώντας, είναι ένας αποτρεπτικός νόμος, ένα, κάτι το οποίο δεν έχουμε ε, δει αλλού, υπά, δεν υπάρχει διαδικασία ένστασης ε, κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει, αντικειμενικά μιλώντας. Δεδομένων αυτών, λοιπόν, μπορείτε μακροπρόθεσμα να πείτε ότι θα γίνει κάτι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πληγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ασμάνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ε, και έκανα μία ερώτηση στον Έλληνα Υπουργό. Του είπα ότι τέσσερα χρόνια αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, ότι ε, τα καταφύγια και εγκαταστάσεις ε, στα ελληνικά νησιά έχουν πρόβλημα, ότι οι διαδικασίες της ασύλου καθυστερούν πάρα πολύ. Βέβαια, υπήρχε στήριξη και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη προς την Ελλάδα Μάλιστα, η ελληνική πλευρά αρνήθηκε τη στήριξη ορισμένων έκρατων μελών και πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι ε, είναι εύκολο να κατηγορούμε την Τουρκία. Αλλά το 2015, όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, ήταν μία λύση αυτό. Τώρα, ε, συμφωνώ για το ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απέσια. Πρέπει πράγματι να γίνει κάτι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Και ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να παροτρύνουμε τις ελληνικές αρχές για να βελτιώσουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρκαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσε όλες οι ερωτήσεις που έγιναν. Νομίζω από το 2015 έχω πάει 10 φορές στη Λέσβο και αναρωτιέμαι αν έχει οποιοδήποτε νόημα να ξανακάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση, ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί. Πραγματικά υπάρχουν παιδιά που περνάνε το χειμώνα σε ε, σκηνές τις οποίες χρησιμοποιούν ε, οι άνθρωποι κανονικά το καλοκαίρι. Υπάρχουν ε, υπαρκτοί κίνδυνοι πυρκαγιάς από, τις από τους αυτοσχέδιους τρόπους ε, θέρμανσης. Υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Υπάρχουν ε, παροχές ε, από εθελοντές. Το 70% ε, της βοήθειας παρέχεται από εθελογές, ε, εθελοντές. Υπάρχει περιθώριο λοιπόν βελτίωσης. Θα συνεχίσουμε να αφήσουμε τους ανθρώπους να υποφέρουν έτσι. Γιατί θα λειτουργήσει αυτό ως αποτρεπτικό μέτρο έτσι ώστε να μην έρθουν άλλοι. Δεν θέλω να κάνουμε συνέχεια τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά να δώσουμε απαντήσεις. Κύριε Σουρμπάνη. Ευχαριστώ. Εγώ πριν από ένα μήνα περίπου ήμουν στη Μόρια, στη Λέσβο και συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση όμω είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κλείσει τη Μόρια. Θα κλείσει τα υπόλοιπα κίτ που έχουμε στα ελληνικά νησιά. Ποια θα είναι η απάντηση μπροστά σε αυτή την καταπήγουσα κατάσταση που δεν είναι κάτι καινούριο θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Τι αποτέλεσμα είχε η νομοθεσία σε σχέση με την πρόσβαση στην υγεία για το θέμα της κάρτας υγείας και επίσης ε, τι ε, έχει γίνει με αυτή την ε, περιστολή των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν εντός των καταβλισμών και τι αποτέλεσμα είχε ε, όταν εστάλησαν ε, ε, τα ΜΑΤ στη Μόρια σε ένα πληθυσμό που έχει τουλάχιστον 3.000 ανηλίκους. Και υπάρχει κατηγορία στο, κατά του ΡΕΑΣΟ ότι αρνούνται να δώσουν συγκεκριμένα χαρτιά σε Ιρακινούς και σε Σύρους. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Ρουίς Δεβέσα. Θέλω καταρχήν να σας επισημάνω κάτι που έχει να κάνει με τις συνθήκες ε, στα hot spot κατά το χειμώνα. Πιστεύω ότι όλοι είδαμε ότι ήδη έχουν περάσει πολλοί χειμώνες υπό αυτές τις συνθήκες και δεν είναι αποδεκτό να επαναλαμβάνονται πράγματα που έχουμε δει στο παρελθόν. Αν υπάρξει και πάλι κάποια αρνητική εξέλιξη, αυτό το χειμώνα θα είναι και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για το θέμα της ε, μεταφοράς, ε, της εκένωσης. Ε, δεν μιλάμε μόνο για τη μεταφορά των ανθρώπων στην υπηρετική χώρα, αλλά μιλάμε και για το θέμα της ανακατανομής των ανθρώπων μεταφέρονται από τα νησιά στο σύνολο των κρατών μιλών και σε καλές συνθήκες, κυρίως όταν μιλάμε για ανηλίκους. Σε σχέση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Υπόθηκε και από τους γιατρούς χωρίς σύνορα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να είναι κάτι ε, περισσότερο θα τονίζεται περισσότερο συμφωνία και θα πρέπει να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο σε οποιαδήποτε αναθεώρηση, δηλαδή σε αντίθεση με το τι έγινε με την αρχική υπογραφή τη συμφωνία με την Τουρκία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε προσπαθώ να μπω στη θέση ορισμένων ε, που μένουν σε αυτά ε, τα στρατόπεδα, αυτούς τους καταβλισμούς. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί μετά από τόσες συζητήσεις, τόση πυρογνωμοσύνη, τα πράγματα χειροτερεύουν. Γίνεται εσκεμμένα έτσι ώστε να τους αποτρελάνουμε και να τα μαζέψουν, να σηκωθούν, να φύγουν ή νομίζουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα έτσι και ότι θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Νομίζω πως ε, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά στηρίζω την έκκληση που γίνεται για άμεση εκένωση. Το θέμα είναι πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και όσο διεξάγονται οι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Συμβουλίου τη Ευρώπη, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρουν μια στέγη. Το θέμα βέβαια είναι να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του προβλήματο και να ξανακοιτάξουμε τη την δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Τα hot spot βέβαια είναι κομμάτι του προβλήματος. Είναι μια προσωρινή ε, λύση, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Το έχουμε δει και στην Ιρλανδία. Μας μιλάνε για προσωρινές λύσεις εδώ και 20 χρόνια, αλλά τίποτα μονιμότερο του προσωρινού. Πρέπει να φροντίσουμε για τους πρόσφυγες. Το κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι αυτή, διότι όλα τα άλλα είναι υποκρισίες. Ε, μας... Ε, λένε για τζιχαντιστές, ε, για προβλήματα και από την άλλη εμεί τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα αίτια τη προσφυγιάς, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις και δεν μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν σπίτια τους, ε, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κάεν. Κοιτάξτε, Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα κάπως, ήμουν σε μια άλλη εκδήλωση. Ευχαριστώ τους ε, παρουσιαστές και τους γιατρούς χωρίς σύνορα που όπως και όλους τους φορείς, τους ε, ΜΚΟ και τους ε, εθελοντικούς οργανισμούς που καλύπτουν διάφορα κενά. Κυρία εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη ΣΑΜΟ ήμουν την περασμένη εβδομάδα. Πού πήγανε τα λεφτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βοήθεια για την Ελλάδα. Διερωτώ με, μπορούμε να έχουμε ένα επίσημο έγγραφο διαφανές όσον αφορά τι δαπάνε που συνδέονται με την καταβολή αυτών των χρημάτων. Δεύτερον, τι θα κάνετε για τη βελτίωση συγκεκριμένα και αμέσω στην κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Υπάρχει τεράστια ευθύνη εκεί και χρηματοδοτούμε πράγματα που δεν ανήκουν στι προδιαγραφέ τη υπαρξαρμοντία πρόσφυγε. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ποια εναλλακτική προτείνεται λοιπόν και τέλο, τι θα κάνετε να βιώσετε την προθεσμία αναμονή ε, για, την, ε, για να εξεταστεί ένα αίτημα ασύλου. Λοιπόν, Στρέφομαι στα μέλη του πάνελ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Περάσαμε το χρονικό όριο και πολλοί από εμά έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Παρακαλώ να το πολύ πέντε λεπτά ο καθένας. Εδώ σταματάμε τη διερμηνία, ε, πέρασε ο χρόνος. Σας ευχόμεθα καλή όρεξη. Γεια σας. Just